Πρέπει να ξεκινήσουμε. Ίσως θα μπορούσατε να χαμηλώσετε λιγάκι τον τόνο των συνομιλιών. Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen. Όπως έλεγα λοιπόν, σας καλωσορίζω στην ακρόαση της υποψηφίας Επιτρόπου για τα ψηφιακά θέματα της κυρίας Νέλη Κρούζ. Καλώς ήρθατε κυρία Κρούζ στην Επιτροπή Βιομηχανίας. Επίσης θέλω να καλωσορίσω τους εκπροσώπους της Επιτροπής πολιτισμού και τους ε, εκπροσώπους της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και της Νομικής Επιτροπής. Έχουμε λοιπόν και άλλα μέλη επιτροπών που δεν είναι της Επιτροπής Βιομηχανίας που ενδιαφέρονται για τα θέματα αυτά και θα προσθέσουν και τα δικά τους ερωτήματα. Θέλω να υπενθυμίσω και πάλι, παρά το γεγονό ότι το έχετε ακούσει πολλές φορές, για το πώ γίνεται η διεξαγωγή τη ακρόαση, 10 λεπτά για την αρχική παρέμβαση τη υποψηφία επιτρόπου, στη συνέχεια θα τεθούν ερωτήματα. Ένα λεπτό για την ερώτηση, δύο λεπτά για την απάντηση, μισό λεπτό για την ε, συμπληρωματική ε, ερώτηση και 1,5 λεπτό για την απάντηση. Ζητώ την κατανόησή σας για το γεγονός ότι είμαι υποχρεωμένος να κρατήσω αυστηρά αυτό το χρονικό διάστημα ώστε να διατηρήσουμε το χρόνο της ακρόασης και να μπορέσουν οι συνάδελφοι που είναι στο τέλος του καταλόγου να θέσουν και αυτοί τις ερωτήσεις τους. Σας ζητώ λοιπόν να είσαστε επακριβείς στην τήρηση του χρόνου ομιλίας και εάν χρειαστεί θα δώσω ένα διακριτικό χτύπημα με το σφυρί στο μικρόφωνο κοντά στο κεφάλι σας για να σας προειδοποιήσω. Νομίζω ότι τα υπόλοιπα είναι ήδη λεχθέντα και γνωστά για όλους σας. Βλέπω ότι είναι κάπως πιο αραιές οι τάξεις μας σήμερα. Ελπίζω ότι βρίσκονται οι συνάδελφοι σε άλλες επιτροπές. Κυρία Κρούς, θα ήθελα τώρα να σας δώσω το λόγο και <clears throat> σας προσκαλώ να κάνετε τις εισαγωγικές σας παρατηρήσεις. Οι συνάδελφοι έχουν ήδη τις απαντήσεις σας, τις γραπτές στο ερωτηματολόγιο και έχετε το λόγο για να παρουσιάσετε τη, τα αρχικά σας σχόλια. Thank you, Chairman And, uh, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αξιότιμα μέλη του Κοινοβουλίου, σας ευχαριστώ για αυτή τη δυνατότητα που μου δίνετε να περιγράψω τις ιδέες μου και να μιλήσω και στους πολλούς Ευρωπαίους που παρακολουθούν αυτή την ακρόαση ζωντανά στους υπολογιστές τους. Η μετάδοση μέσω διαδικτύου, το web streaming, είναι ένα πολύ ισχυρό σύμβολο διότι συμβολίζει πόσο σημαντική είναι η τεχνολογία της ενημέρωσης και της πληροφορικής που έχει φτάσει έχει τόσο μεγάλο σημαντικό κομμάτι στην ευρωπαϊκή ζωή. Είναι γεγονός ότι κάθε Ευρωπαίος κάθε μέρα βλέπει ότι η τεχνολογία αυτή προωθεί την ανάπτυξη την τεχνολογία βελτιώνει την ποιότητα ζωής μας και η τεχνολογία της πληροφορικής συνδέει τις κοινότητές μας. Αυτή η τεχνολογία βελτιώνει την καθημερινή μας ζωή και μας κάνει πιο πλούσιους. Το ψηφιακό πρόγραμμα θα πρέπει να μεγιστοποιήσει αυτά τα αποτελέσματα και αυτά τα κέρδη και αν με υποστηρίξετε και αν με ε, επικυρώσετε ως ε, επίτροπο θα ζητήσω την υποστήριξή σας για να πετύχουμε αυτά τα κέρδη σε όλο το φάσμα των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Έχουμε πάρα πολλές επιτυχίες στον τομέα αυτό, τις τεχνολογίες της πληροφορικής, των πληροφοριών, αλλά πάντα καταφέρουμε καλύτερα. Δεν μπορούμε να είμαστε εφησυχασμένοι, ανταυτού χρειαζόμαστε μια άλλη νοοτροπία που ενστερνίζεται τη δημιουργία νέων αγορών και, ε, και διαβίωσης. Και θα πρέπει να επενδύσουμε έξυπνα για να εκμεταλλευτούμε τα δυνατά μας σημεία και να δημιουργήσουμε τις συνθήκες για την ψηφιακή οικονομία στην Ευρώπη, να την κάνουμε την ψηφιακή οικονομία να ανθίσει. Και αν επικυρωθεί ο διορισμός μου ως επίτροπος για, την ψηφιακή, για το ψηφιακό πρόγραμμα, θα προσπαθήσω να δημιουργήσω ένα περιβάλλον στο οποίο θα δημιουργηθούν οι νέες Nokia, τα νέα Skype και οι νέες προδιαγραφές για τα κινητά τηλέφωνα. Έχοντας το σωστό πρόγραμμα τώρα, ετοιμάζοντάς το, θα συμβάλλουμε σε μια γενιά ανάπτυξης και απασχόλησης στην ε, Ευρώπη. Κατά την άποψή μου υπάρχουν έξι οικοδομικοί λύθοι για να πραγματοποιήσουμε το πρόγραμμα. Πρώτα απ' όλα έχουμε καινοτομία και έρευνα. Μεγαλύτερη δέσμευση για να διεξαχθεί, να πραγματοποιηθεί έρευνα και καινοτομία και περίπου 1,7 δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο για κοινοτική έρευνα και ανάπτυξη και καινοτομία. Για τον τομέα αυτό. Ε, είναι σημαντικό ποσό για τον τομέα αυτό που συζητούμε, για την τεχνολογία της πληροφορικής, των πληροφοριών. Αυτό είναι λιγότερο όμως από το ποσό που διαθέτει κάθε χρόνο για έρευνα και ανάπτυξη το Google. Άρα δεν μπορούμε να σπαταλήσουμε ούτε ένα ευρώ θα πρέπει τα χρήματα αυτά να χρηματοδοτήσουν την έρευνα και ανάπτυξη που δεν θα γινόταν χωρίς αυτά τα ποσά και θα πρέπει να τα προωθήσουμε όλα αυτά όσο δυνατόν περισσότερες ιδιωτικές και εθνικές επενδύσεις γίνεται και θα πρέπει να βασιστούμε στα ταλέντα των ερευνητών μας ούτω ώστε να δημιουργήσουμε ένα νέο οικοσύστημα όπου οι εταιρείε της πληροφορικής οι ευρωπαϊκές όλων των μεγεθών να μπορούν να παράγουν ε, πάρα πολύ ποιοτικά προϊόντα που να σταθούν στην παγκόσμια αγορά. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα προγράμματα πλαίσια, τα παραδοσιακά τους μέσα για πετύχοντα σκοπό ή να χρησιμοποιήσουμε σκοπό ή να χρησιμοποιήσουμε διάφορες μορφές συνεργασίας ιδιωτικού δημόσιου τομέα ή ε, διάθεση, πώληση, προδιαθέσεως στην αγορά. Θα πρέπει ε, η τεχνολογία να βελτιώνει τη ζωή η τεχνολογία που θα επιτρέπει στους πιο ηλικιωμένους Ευρωπαίους να ζουν ανεξάρτητα, ε, τεχνολογίες που μειώνουν το κόστος της υγειονομικής περίθαλψης, με εντυπωσιάζει η Δανία με αυτά που κάνει, είχαν ένα έξοχο άρθρο η New York Times πάνω σε αυτό, που έδειχναν ότι ηγείται η Δανία σε αυτό το τομέα, ε, περνάει και κατά πολύ τις Ηνωμένε Πολιτείες, δίκτυα που συνδέουν ανθρώπους και επιχειρήσεις, με πιο και νοτόμους τρόπους, τεχνολογία που κάνει πιο πράσινη, πράσινες τις μεταφορές και πιο ασφαλής Δεύτερος οικοδομικός λήθος, οι υποδομές. Οι πολίτες και επιχειρήσεις όλο και περισσότερο θα πρέπει να συνδέονται ανα πάσα στιγμή οπουδήποτε. Ε, και για να συμβεί αυτό θα πρέπει να επενδύσουμε σε διευρωπαϊκά βριζονικά δίκτυα και ασύρματες εφαρμογές που χρησιμοποιούν το ε, ραδιοφωνικό φάσμα αποτελεσματικά. Και αυτό απαιτεί κατάλληλα κίνητρα για να τονωθεί ιδιωτική επένδυση χωρίς να ξαναμιγηθούν μονοπόλια στα δίκτυα. Και θα πρέπει οι επενδύσεις οι κρατικές να έχουν συγκεκριμένους στόχους που βελτιώνουν τη λειτουργία της αγοράς. Και με αυτή την υποδομή χρειάζονται ανταγωνιστικές αγορές, ώστε οι υπηρεσίες επικοινωνιών να είναι διαθέσιμες και σε καλές τιμές, δίκαιες τιμές. Τρίτος οικοδομικός λίθος. εμπιστοσύνη και ασφάλεια. Η τεχνολογία αυτή, η ψηφιακή, θα πρέπει να είναι αντικείμενο εμπιστοσύνη. Αν φοβούνται οι Ευρωπαίοι για την ιδιωτική τους σφαίρα, φοβούνται για απάτες ή ανησυχούν για απειλές κατά των παιδιών τους, τότε θέτουμε τροχοπέδι στην ψηφιακή τεχνολογία και θα πρέπει να εμπιστευόμαστε τον δημόσιο έλεγχο για την διαχείριση του διαδικτύου. Τέταρτος οικοδομικός λήθος πρέπει να υπάρχει δικαιοσύνη. Για να είμαστε δίκαιοι και ανταγωνιστικοί, οι πολίτες και οι επιχειρήσεις πρέπει να έχουν την πρόσβαση και τις δεξιότητες, ούτως ώστε να αποφεληθούν από αυτή την τεχνολογία. Δεν είναι τίποτα ψηφιακή τεχνολογία, μα λησμονούμε τους ανθρώπους και μπορούμε να δημιουργήσουμε δίκτυα και συσκευές αλλά αν οι πιο ηλικιωμένοι και οι πιο μειονεκτούντες Ευρωπαίοι δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν όλα αυτά, οι επιχειρήσεις δεν μπορούν να βρουν το κατάλληλο προσωπικό με τις δεξιότητες, δεν πετυχαίνουμε τους στόχους μας. Πέμπτος οικοδομικός λήθος, ψηφιακή κοινωνία. Αυτή εξαρτάται από ανοιχτά πρότυπα και διαλειτουργικότητα. Και με αυτό υπόψη μας οι δημόσιοι φορείς θα πρέπει να ε, κάνουν πράξη τα λόγια τους αν δεν χρησιμοποιούν ανοιχτά πρότυπα, ανοιχτά συστήματα, γιατί να το κάνουν οι πολίτες. Εγώ θα το επιδιώξω να το πετύχω από τοπικό επίπεδο μέχρι ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Ε, τέτοια στοιχεία όπως χάρτες, ο καιρός, πληροφορίες για την υγεία δεν καλύπτονται από διαλειτουργικότητα, πώς μπορούν να χρησιμοποιηθούν με καινούριου τρόπους. Και θέλω να διερευνήσω νέους τρόπους για να αναπτύξουμε τα πρότυπα για την ψυχιακή τεχνολογία στην ε, Ευρώπη. Έκτος οικοδομικός λήθος, ε, ενιαία αγορά σε απευθεία σύνδεση online. Η ευρωπαϊκή μας αγορά στο διαδίκτυο είναι ε, ένα σύνολο εθνικών αγορών και το λέω και κομψά όλα. Είναι διρεμένη αυτή η αγορά με διαφορετικές ρυθμίσεις και δημιουργεί ένα σύστημα που απογοητεύει τους καταναλωτές και περιορίζει τις επιχειρήσεις. Και θέλω να συνεργαστώ μαζί σας, εάν επικυρώσετε το διορισμό μου ως Επίτροπο, θα συνεργαστώ μαζί σας, τα κράτη-μέλη και τους συναδέλφους στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να προωθήσουμε, να πολεμήσουμε για μια πραγματική ενία αγορά ηλεκτρονική, online, για αγαθά, υλικά και πολιτιστικά και διάφορες υπηρεσίες που δεν μπορούμε καν να φανταστούμε. Έχουμε το φυσιακό πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής επ' αυτής της βάσεως. Για να την υλοποιήσουμε θα πρέπει να βασιστώ ε, στην έκθεση ε, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που ετοιμάζει η κυρία Ντελκαστήγιο για την όλη ανάπτυξη που θα ακολουθήσουμε το 2015 ε, θα συμφωνήσετε ότι αυτή η οικοδομική λύθη, αυτά τα κομμάτια είναι μόνο τα μέσα για την επίτευξη του σκοπού είτε μέσω προγράμματος όπως το Ευρωπάνα, Ιστορία ή καλύπτοντας το ψηφιακό χάσμα, όλες αυτές οι προσπάθειες έχουν το ίδιο αποτέλεσμα. Είναι ευρωπαϊκές λύσεις που πετυχαίνουν ευμάρια για όλους τους πολίτες. Καλύτερο επίπεδο διαβίωσης στην καθημερινή ζωή όλων των Ευρωπαίων. Πώς θα εφαρμόσω αυτές τις ιδέες αν επικυρώσετε το διορισμό μου. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα έχει, έχει συμβάλει κατά τα μάλα όσον αφορά την οδηγία για τις τηλεπικοινωνίες και τα απτυτικοστικά μέσα. Θα πρέπει τώρα τις δυνατότητες που υπάρχουν, όπως πολιετή προγραμματισμό φασμάτων, αυτά να τα κάνουμε πρακτικές. Και για να το καταφέρουμε αυτό, νομίζω ότι χρειαζόμαστε στεναρή υποστήριξη των κρατών μελών και σκληρές απαντήσεις όμως έναντι εκείνων που παραβιάζουν ή αγνοούν το κοινοτικό δίκαιο και τις διάφορες προθεσμίες για την εφαρμογή των διατάξεων των ευρωπαϊκών. Αν με υποστηρίξετε, έχω τη φιλοδοξία να συνεργαστώ με την βιομηχανία και τους εμπειροβημένους και τους ενδιαφερομένους να καταλήξουμε σε ε, καινοτόμε συνεισφορές για την υλοποίηση αυτού του ψηφιακού προγράμματος. Πρέπει να είναι υποφελές για όλους το πρόγραμμα διότι νομίζω ότι έτσι μπορούμε να πετύχουμε τα βέλτιστα αποτελέσματα. Σας διαβεβαιώνω, εάν αυτό δεν οδηγήσει σε λύσεις, οι δημόσιες αρχές θα πρέπει να υπομισθούν τις ευθύνες τους, ε, ούτω ώστε να μπορέσουμε να πετύχουμε τους ε, κοινούς μας στόχους. Εν τέλει, θα ήθελα να αναφέρω τι με οδηγεί στον να ενδιαφέρομαι τόσο πολύ για αυτό το χαρτοφυλάκιο. Εγώ ενθουσιάζομαι με την προπτική να αντιμετωπίσω το θέμα αυτής τη ψηφιακή ατζέντα αυτού του προγράμματος και σαν επίτροπος για τον ανταγωνισμό έχω καλό ιστορικό φέροντα συναθρίζοντας κόσμο κάνοντα συστήματα να λειτουργήσουν και αυτό βέβαια δεν δημιουργεί μόνο φίλου, δεν να σα το πω, αλλά ξέρει ο κόσμος ότι είμαι ευθύ, είμαι διαφανής και ακολουθώ μια γραμμή για να πετύχω αποτελέσματα για τους λαούς στην Ευρώπη. Συναφρίζοντας ανθρώπους, ενώντας ανθρώπους, κάνοντας πράγματα όσον αφορά τη διαλειτουργικότητα, τα ανοιχτά πρότυπα ε, για τα τέλη που πληρώνουν καταναλωτές, για την ευρωζωνική αγορά, για τις εκπομπές, για την αγορά σε απευθεία σύνδεση με το διαδίκτυο, βοηθάω και τους πολίτες και τις επιχειρήσεις ε, και τους εντάσσω στις ευθύνες μου και δημιουργώντας οι ιδέες που βοηθούν την υλοποίηση του προγράμματος. Ε, κάνοντας όλα αυτά θα σας δείξω ότι μπορώ να τα κάνω. Αυτό είναι το όραμά μου για το ψηφιακό μέλλον. Τώρα θα ήθελα να ακούσω και ποιες είναι οι συμβουλές σας. Θα επιδιώξω βέβαια τις συμβουλές σας και την υποστήριξή σας αν επικυρωθώ στη θέση μου και θα επιδιώξω να έχουμε στενή συνεργασία. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, κυρία Ντελκαστίγιο. Έχει το πρώτο ερώτημα. Ευχαριστώ πολύ κυρία. Κύριε Πρόεδρε, κυρία Υποψήφια Επίτροπε, κυρία Κρούς, εξ της πολιτικής μου ομάδος, θέλω να σας καλωσορίσω στην ε, ακρόαση αυτή. Ο πρόεδρος Μπαρός, όπως γνωρίζετε πολύ καλά, έχει διαδηλώσει το πολιτικό του πρόγραμμα για την επόμενη Κομισιόν και τόνισε ότι περιλαμβάνει μια ευρωπαϊκή ψηφιακή ατζέντα. Καταρχήν να ξεπεράσουμε τα εμπόδια για τη δημιουργία μιας ενιαίας ανοιχτής και ανταγωνιστικής ψηφιακής αγοράς, να προωθήσουμε τις επενδύσεις στις συνδέσεις υψηλής ταχύτητος και επίσης να αποφύγουμε κάθε μορφή ψηφιακού χάσματος. Προφανώς το Κοινοβούλιο μας θα συζητήσει τα θέματα αυτά στις αρχές Φεβρουαρίου. Την ε, έκθεση αυτή, τη δική μου, για την ψηφιακή ατζέντα. Είναι γεγονό ότι η σωστή λειτουργία τη ψηφιακή οικονομία θα είναι απαραίτητη για την καλή λειτουργία όλη τη Ευρωπαϊκή οικονομία. Παρ' όλα αυτά γνωρίζουμε όλοι ότι απέχουμε ακόμα πολύ από το να μπορέσουμε να επιτύχουμε στην Ευρώπη μια πλήρη λειτουργία μια πλήρου και ενιαίας αγορά σε ό,τι αφορά τι διαδικτυακέ υπηρεσίε. Απέχουμε πόρο όπω δείχνουν και τα στοιχεία. Μόνο το 7% των συναλλαγών που γίνονται μέσω του διαδικτύου γίνονται από καταναλωτές με διαμεθοριακό χαρακτήρα. Μόνο 7% λοιπόν διαμεθοριακές διαδικτυακές συναλλαγές. Έχουν ανακοινωθεί πολλά μέτρα, αλλά πιο συγκεκριμένα ποια είναι τα μέτρα προτεραιότητος τα οποία με κατεπίγοντα τρόπο θα προτείνετε εσείς για να επιτευχθεί αυτή η ενιαία και μοναδική ψηφιακή αγορά. Κυρία Κύριε Πρόεδρε, όπως ε, τόνισε η κυρία Βουλευτής, το θέμα αυτό είναι ένα θέμα μεγάλης προτεραιότητος, όχι μόνο για τον πρόεδρο Μπαρόσο, αλλά σας διαβεβαιώ για όλους τους εμπλεκόμενους στην δυνητική, ε, στο δυνητικό αυτό σχήμα της νέας Κομισιόν. Όταν μιλάμε για την ψηφιακή ατζέντα, θα ήθελα να κάνω δύο παρατήρησεις που έρθω ακριβώ στο ερώτημά σας εάν μιλάμε για την ψηφιακή ατζέντα, αυτό δεν είναι αυτός σκοπός. Είναι ένας, ένα εργαλείο για να μπορέσουμε τελικά να καταλάξουμε σε μια διαφορετική Ευρώπη. Οι τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας δίνουν σημαντικές βελτιώσεις στην καθημερινή μας ζωή. Μιλάμε για τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις επιχειρήσεις. Θέσεις εργασίας, ευμάρεια, ποιότητα ζωής, η δυνατότητα να επικοινωνούμε. Νομίζω λοιπόν ότι εδώ υπάρχουν κάποιες προτεραιότητες οι οποίες είναι πολύ σημαντικές. Χρειάζεται να επιτύχουμε μια ενιαία αγορά στον ψηφιακό τομέα και ακριβώς εδώ μιλάμε για το δημιουργικό περιεχόμενο στο διαδίκτυο, εκεί πρέπει να υπάρχει μια ενιαία αγορά. Θα υπάρξει λοιπόν μεγάλη διαφορά αν το επιτύχουμε αυτό. Αυτό το οποίο εγώ έκανα ως Επίτροπος Ανταγωνισμού ήταν να προσπαθήσω να συνενώσω. Πιστεύω τα γνωρίζετε αυτά για την ψηφιακή ενιαία αγορά στην περίπτωση της στρογγυλής τραπέζης για τα διαδικτυακά θέματα και αυτό ήταν ανάληψη κινδύνου να έλθουν και να συναντηθούν σε μια στρογγυλή τράπεζα εταίροι και παίκτες οι οποίοι συνήθως συναντιόντουσαν στα δικαστήρια. Ήταν ένα μεγάλο ρίσκο λοιπόν, αλλά ο στόχος ήταν να καταλήξουμε σε ένα έγγραφο προβληματισμού σε σχέση με το περιεχόμενο σε μια ενιαία αγορά ψηφιακών προϊόντων. Και νομίζω ότι είναι πολύ ενδιαφέρουσα και για σας αυτή η πρωτοβουλία και η δημόσια διαβούλευση η οποία έχει ξεκινήσει για να μπορέσουμε να ξεπεράσουμε τους εδαφικούς περιορισμούς στην αδειοδότηση του δημιουργικού περιεχομένου και όλος αυτός ο προβληματισμός έχει σαν στόχο να καταλήξουμε σε καλύτερο περιεχόμενο και μεγαλύτερη προστασία για τους πνευματικούς δημιουργούς. Μαζί με τον Μισελ Μπαρνιέ, λοιπόν, έχω σαν στόχο να προχωρήσω προς αυτή την κατεύθυνση προτεραιοτήτων και όχι απλώς να μιλάω γενικόλογα. Eh, Ευχαριστώ. Δεύτερη και σύντομη ερώτηση. Μέσα σε αυτό το ρυθμιστικό πλαίσιο είναι εγγενής και η ιδέα του να μειώσουμε την εκ των προτέρων ρύθμιση, την εξάντε ρύθμιση στα πλαίσια αυτά τα ψηφιακά για να λειτουργήσει πλήρως ο ανταγωνισμός. Στην αγορά επικοινωνιών έχουμε κάνει τηλεπικοινωνία, έχουμε φέρει πολλά καινοτόμα στοιχεία τα οποία προωθούν τον ανταγωνισμό. Αν λάβουμε υπόψη το δικό σα παρελθόν ω επιτρόπου ανταγωνισμού, Πώ πιστεύετε ότι θα μπορέσετε να επιτύχετε την σταδιακή μείωση τη εκ των προτέρων ρύθμιση και επίση θεωρείτε ότι η απόλυτη άρση κάθε εκ των προτέρων ρύθμισης μπορεί να είναι κάτι το εφικτό κατά τη διάρκεια της θητείας σας. Αν είναι πέντε χρόνια, ναι. Σας ευχαριστώ. Η ε, κυρία Τράτμαν. Merci, Monsieur le Président. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Κυρία Κρός, ξέρετε όπως και εμείς τον κινητήριο ρόλο που πρέπει να παίξει η ψηφιακή τεχνολογία για την ανάκαμψη την οικονομική και την κοινωνική της Ευρώπης. Η ομάδα μου θέλει να σας ακούσει και να ακούσει ποιε είναι δεσμεύσει σα, ποια είναι η βούλησή σα, ούτω ώστε σε ευρωπαϊκή κλίμακα να εφαρμοστεί μια πραγματική βιομηχανική πολιτική που μέχρι τώρα φαινόταν καμία φορά να κάπου να χανόταν μέσα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πώ μπορεί να εφαρμοστεί μια τέτοια πολιτική που είναι αποτελεσματική όσον αφορά την επένδυση σε δίκτυα, δημιουργεί θέσει απασχόληση και επιτρέπει καινοτόμε και φθηνέ ε, υπηρεσίε για του καταναλωτέ. Ακούσαμε τον κύριο, τον κύριο Κουίν, με τον οποίο έχετε ευθύνε, μερίζεστε τι ευθύνε όσον αφορά την ανταγωνιστικότητα. Έχετε κοινό όραμα όσον αφορά αυτό το θέμα. Οι σχέσει με τη Γενική Διεύθυνση αυτή, ε, πώ θα συνδυαστεί για την ανταγωνιστικότητα. Θέλουμε ένα σαφέ μήνυμα από εσά και συγκεκριμένε ε, δεσμεύσει. Κυρία Κρούς, σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η αξιότιμη βουλευτής με ρωτάει αν υποστηρίζω μία προσέγγιση βιομηχανικής πολιτικής. Είμαι απόλυτα βέβαιη ότι με γνωρίζετε εντωμεταξύ λίγο καλύτερα. Είμαι πολύ ρεαλίστρια. Δεν θα μπορούσα να είμαι πιο Ολλανδέζα από την άποψη αυτή. Και ανυπομονώ να επιλύσουν τα θέματα αυτά. Να εξηγήσω λοιπόν με την ευκαιρία αυτή το εξή. Αν εγκριθώ στη θέση μου, αν μου δοθεί η ευκαιρία να συμπληρώσω όσα χρειάζονται στην ψηφιακή ατζέντα, να αναφέρω για παράδειγμα τα NGAs, και όσα χρειάζονται για να γίνουν οι νέες επενδύσεις στις νέες αυτές οι υποδομές. Εμείς λέμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι χρειάζεται 100% ευρυζωνική κάλυψη. Δεν χρειάζεται πολύ φαντασία για να καταλάβει κανείς ότι πρέπει πραγματικά να αρχίσουμε αύριο, κατεπηγόντως. Ιδάλλως δεν πρόκειται να πετύχουμε τους στόχους μας. Αν αυτό εννοείται μιλώντας για βιομηχανική πολιτική, ναι, συμφωνώ, να πω. Αλλά για μένα είναι πολύ σημαντικό να πληρώσουμε, να καλύψουμε για να σοβαρευτούμε. Νομίζω ότι μιλώντας για αυτό το τμήμα της ψηφιακής ατζέντα, για τη συνολική προσέγγιση της 100% ευρυζωνικής κάλυψης στην Ευρώπη, θα πρέπει να τράξουμε την ευκαιρία αυτή για δύο λόγους. Κατά πρώτον, όντως συμπληρώνει την ανταγωνιστικότητά μας αυτό, την ευκαιρία μας να προηγηθούμε στον κλάδο αυτό, αλλά παράλληλα αποτελεί και μια εξαιρετική ευκαιρία για να δώσουμε μια όθηση στην οικονομική ανάπτυξη, να δημιουργήσουμε θέσεις εργασίας και τα χρειάζεται να σας εξηγήσω ότι αυτό δεν είναι κάτι το οποίο Χρειάζεται να περιμένουμε για να ξεκινήσουμε. Και μιλάμε για μια πολιτική για τη δημιουργία θέσεων εργασία και για την πρόθεση της οικονομίας. Κύριε suis... Ναι, δεν είμαι απόλυτα φίλη σα, γιατί δεν έχω ικανοποιηθεί ιδιαίτερα από την απάντησή σας. Ιδίω στο τμήμα το οποίο αφορά την καινοτομία. Θέλω να σα θέσω το εξή θέμα. Οι πολίτε περιμένουν από τις αρχέ να σεβαστούν τα θεμελιώδη δικαιώματά σας. Γνωρίζετε τις συζητήσεις οι οποίες έχουν λάβει η χώρα μέσα στα πλαίσια του πακέτου τηλεπικοινωνιών στην, σε ό,τι αφορά το ρόλο του ίντερνετ για την, προστασία, για την ε, ελευθερία έκφρασης αλλά και την προστασία των ιδιωτικών δεδομένων και της ιδιωτικής ζωή Πώ μπορείτε να εξασφαλίσετε ότι η συμβαστική λύση δεν θα αλλοιωθεί στην <clears throat> εφαρμογή της ή θα τροποποιηθεί από μια παγκόσμια συμφωνία όπως η Άκτα, η οποία αυτή τη στιγμή είναι υποδιαπραγμάτευση από τη Γενική ε, Διεύθυνση της Κομισιόν, η οποία είναι αρμόδια. Μαζί με την κυρία Ρέντινγκ, λοιπόν, θα είσαστε μια ομάδα κρούσης για να επιτύχετε αυτά τα πράγματα ή όχι. Δεν χρειαζόμαστε... Δεν χρειάζομαι πολύ χρόνο να σας υπενθυμίσω ότι εγώ υποστηρίζω πάρα πολύ αυτήν την ε, αντιμετώπιση και για μένα το ίντερνετ είναι ένα θεμελιώδες δικαίωμα και αν μιλάτε για τη συμφωνία η οποία έχει γίνει για την μη εφαρμογή αντιμέτρων Έχω συζητήσει αυτό το θέμα και με τον Κάρελ Ντεχούχτ, ο οποίο είναι υπεύθυνο για το εμπόριο. Και ο στόχο των διαπραγματεύσεων άξα, όπω γνωρίζετε, είναι να μπορέσουμε να καταλήξουμε σε ένα διεθνέ πλαίσιο το οποίο θα ε, εφαρμόσει ένα γενικό πλαίσιο κατά τη ε, κυκλοφορία παραποιημένων προϊόντων και για τη διατήρηση των κανόνων του copyright με ένα κοινό τρόπο αντιμετώπιση αυτών των παραποίησεων που γίνονται πολλέ φορέ από εγκληματικέ οργανώσει Και από αυτή την άποψη και μέσα στη διαδικασία διαπραγματεύσεων της ΑΚΤΑ οι διαπραγματεύοντες εταίροι πρέπει να αντιμετωπίζουν και την αυξανόμενη σημασία του ίντερνετ. Δεν υπάρχει κάποιο κείμενο το οποίο έχει τη συμφωνία μέχρι στιγμή. Έχει υπάρξει ένα πρώτο, μια πρώτη πρόταση από τις ΗΠΑ. Για μας όμως το σημαντικό είναι οι διεθνείς εταίροι μας να εγγυηθούν καταρχήν το ίδιο επίπεδο προστασίας διεθνών πνευματικών δικαιωμάτων που εφαρμόζει αυτή τη στιγμή η Ευρωπαϊκή Ένωση μαζί με όλες τις εγγυήσεις του κοινοτικού κεκτημένου. Και νομίζω και ο Κάρλ Φανγκούχτ θα σας πει το ίδιο πράγμα, ότι αυτές είναι εγγυήσεις που χρειαζόμαστε. Η Κομισιόν συμφωνεί με το τωρινό επίπεδο εναρμόνισης των πνευματικών, εναρμόνισης των πνευματικών δικαιωμάτων και δεν θα υπάρξει μεσοκιακόπορτας άλλη μορφή ε, εναρμόνισης. Θα πρέπει λοιπόν οι άλλοι να προσεγγίσουν τη δική μας θέση. Η κυρία Έξα, παρακαλώ πάρα πολύ να είσαστε πιο προσεκτικοί για τον χρόνο, κυρία Κρούς. Δεν θα ήθελα να σας διακόπτω, αλλά μου δημιουργεί δυσκολίες αν πρέπει να το πράττω. Κυρία Εκ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καταρχάς θα ήθελα εξ της ομάδας μου να σας καλωσορίσω στην ακρόαση αυτή, κυρία Κρούς. Το διαδίκτυο αποτελεί ένα εξαιρετικό όργανο για την κοινοτομία και την πρόοδο. Και χάρη στο γεγονό ότι έχουμε την ελευθερία να κάνουμε ο καθένα τι δικέ μα επιλογέ. Αλλά αυτό οδηγεί σε ορισμένε περιπτώσει σε απόπειρε ελέγχου του διαδικτύου από το κράτο. Για παράδειγμα, στην Κίνα με το πακέτο τηλεπικοινωνιών που εγκρίθηκε το φθινόπωρο καταδείξαμε στην Ευρώπη ότι υπάρχει η δυνατότητα να υπάρχει νομική βεβαιότητα για τους πολίτες με τον κατάλληλο τρόπο. Θα ακολουθήσετε αυτό τον δρόμο που έχει χαράξει η Ευρώπη για να εγγυηθείτε την ουδετερότητα του δικτύου και να μην επικρατήσουν ε, κράτη, για παράδειγμα, στον έλεγχο του δικτύου. Η κυρία Κρούς, απάντηση είμαι υπέρ. Και σε αυτό με βρίσκεται, σύμφωνη και αυτό φαντάζομαι ότι σας βρίσκει και όλους τους υπόλοιπους ε, σύμφωνους ότι η ουδετερότητα του δικτύου θα πρέπει να είναι προσωπικό θέμα. Και με επασχολεί ιδιαίτερα αυτό το θέμα. Είναι λοιπόν εξαιρετικά σημαντικό και από πλευρά Ευρωπαϊκή Επιτροπή να διατηρήσει τον ουδέτερο χαρακτήρα του δικτύου, αλλά υπάρχουν, υπάρχουν κάποιοι λόγοι για τους οποίους θα πρέπει να είμαστε άγρυπνοι για νέες προκλήσεις σε ό,τι αφορά την ουδετερότητα του δικτύου, που μπορούν να προκληθούν από πολλές πηγές. Για παράδειγμα, μέσω των υπηρεσιών VoIP, voice over IP και ε, χρειαζόμαστε διαφάνεια και πάντα αυτό υποστηρίζουμε και γι' αυτό άλλωστε αναθεωρήσαμε και τους κανόνες της τηλεπικοινωνίας για να ενισχύσουμε την ε, διαφάνεια για τους καταναλωτές. Αναφέρατε την περίπτωση της Google στην Κίνα. Νομίζω ότι όλοι συμφωνούμε ότι πρόκειται για μια περίπτωση που αποδεικνύεται ότι υπάρχει υψηλό επίπεδου ε, επιθέσεις στον χώρο. Δεν τίθεται θέμα δηλαδή μη επαγρύπνησης. Είναι πάρα πολύ δημιουργικές αυτές οι επιθέσεις. Και επίσης, και αυτό είναι πολύ ανησυχητικό, αν αποδεχτεί παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των ακτιβιστών μέσω του διαδικτύου. Θα είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Πολύ ανησυχητικό και είναι πολύ σημαντική φυσικά και η ελευθερία της έκφρασης. Άρα με το περιστατικό αυτό καταδεικνύεται ότι κάποια θέματα τα οποία όλοι θεωρούμε δεδομένα θα πρέπει και αυτά να ξαναποδεχτούν. Η συνάδελφος Έκε. Ευχαριστώ. Πολλοί νέοι ανησυχούν ιδιαίτερα για θέματα ακεραιότητας, θέματα δικαίου νεολαία του κόμματό μου στην ε, Σουηδία, για παράδειγμα, στη χώρα μου, συζητάει το θέμα αυτά. Και ο Ευρωπαίος διαμεσολαβητής μπορεί να αποκτήσει επιπλέον αρμοδιότητα στο θέμα αυτό, για θέματα ιδιωτικής σφαίρας και ακεραιότητας. Καταλαβαίνω τι λέτε, αλλά νομίζω ότι δεν νομίζω ότι είναι στο πεδίο των αρμοδιοτήτων του. Αυτός είναι υπεύθυνο για το εσωτερικό της οργάνωσή μας. Νομίζω ότι υπάρχουν κι άλλες, πολλές δυνατότητες, αλλά επιτρέψτε μου να το σκεφτώ και να το συζητήσω αργότερα μαζί σας. Μαζί με εσά και τους συναδέλφους σας, γιατί αυτό αποτελεί ένα βασικό θέμα, αλλά σε συγκεκριμένη περίπτωση δεν ξέρω αν ο διαμεσολαβητής είναι το κατάλληλο άτομο για να επιλύσει το πρόβλημα. Σα ευχαριστώ, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καλώ ήρθατε κυρία Κρυούζαν, ονόμα των Πρασίνων. Εκτιμήσαμε τι υπηρεσίε σα, όταν ήταν επικεφαλή τη Γενική Διευθύνσεω Ανταγωνισμού. Θα θέλαμε να συνεχίσετε, το δείτε, θα στέλνουμε εδώ, αλλά κάνατε έξοχη δουλειά εκεί πέρα. Και νομίζω ότι ο διάδοχό σα θα έχει πολλή δουλειά να κάνει για να φτάσει στο επίπεδό σα, να το κρατήσει το επίπεδο των δράσεών σα. Θα ήθελα να συνεχίσω το θέμα τη ουδετερότητα του δικτύου. Είπα το διαδίκτυο είναι ένα εργαλείο στην υπηρεσία τη αγορά, είναι ένα εργαλείο στην υπηρεσία των δημοσίων υπηρεσιών, αλλά είναι και ένα εργαλείο για τη δημοκρατία. Ένα εργαλείο μέσω του οποίου τα δικαίωμα τη έκφραση, πρόσβαση στην πληροφορία μπορεί να το εγγυηθούμε καλύτερα μέσω αυτού του μέσου παρά μέσω οδήποτε άλλου μέσου. Θα επιβάλλεται την ουδετερότητα του δικτύου. Βεβαίω μπορούμε να δούμε πώ οι διάφοροι πάροχοι θα ελέγχουν την κυκλοφορία ή όχι. Και επίσης τι γίνεται με τη θεματική επιλογή. Κάτι που εμποδίζει την ουδετερότητα του δικτύου. Γνωρίσατε στην περίπτωση Microsoft τα θέματα αυτά. Πώς θα δράσετε στην τεχνολογία, στην ε, τεχνολογική πτυχή της ουδετερότητας του δικτύου ούτω ώστε το δίκτυο, το διαδίκτυο να παραμείνει ουδέτερο. Η κυρία Κρούσε έχει το λόγο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 με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και παρόλα αυτά κάτι κατάφερε να πάει στραβά. Θα αφαιρέσουμε τα λεφτά αυτά από το τέλος. Καταλαβαίνατε και σουηδικά νομίζω. This is just to fill the time. Κάνω αυτό για να περάσει η ώρα. Haben Sie die Frage verstanden, Frau Kruse, eben noch? Καταλάβατε την ερώτηση. I will manage. Θα καταφέρω, θα καταφέρω. Microsoft είπατε και ιδιαιτερότητα του δικτύου η συνέπεια των τεχνολογικών ε, επιλογών σε κλειστέ τεχνολογίε που επηρεάζουν την ιδιωτικότητα του δικτύου. Τι μπορείτε να κάνετε στο νέο σα ρόλο πάνω σε αυτό το θέμα. Απάντηση. Εμείς δεν σταματάμε τις δυνατότητες στην ύπαρξη κάποιων τεχνολογιών. Μιλάτε για ανοιχτή πηγή, open source, ανοιχτό κώδικα θα πρέπει να υπάρχει αυτό, διαφορετικά θα δημιουργείται πρόβλημα δεσπόζουσας θέσης. Κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης, αυτό δεν πρέπει να γίνει. Η ουδετερότητα του δικτύου σημαίνει ανοιχτή και σαφής ουδετερότητα του δικτύου. Για να συμπληρώσω, όσον αφορά το ρόλο που έπαιξε η ψηφιακή τεχνολογία, για να πετύχουμε μια ε, οικονομία των πόρων. Ε, υπάρχουν πολλοί πλειοτικοί τομεί, μεταφορέ, αποδοτικότητα τη ενέργεια, κινητικότητα κλπ. Τι πρωτοβουλίε θα θέλατε να αναλάβετε τόσο ώστε να επιταχύνετε τι συνέπειε τη τεχνολογία αυτή όσον αφορά τη μεταμόρφωση της οικονομίας μας. Απάντηση. Αρκετά πράγματα μπορούμε να κάνουμε σε συνεργασία με πολλού συναδέλφου. και αυτή είναι η ελκυστικότητα του χαρτοφυλακίου δεν είναι κάτι πεπερασμένο, κλειστό. Αναφέρεται στην ηλεκτρονική υγεία μέσω διαδικτύου, ε, πολιτισμό, εμπόριο, οικονομία, ενιαία αγορά, ενέργεια και πώς μέσω πρωτοβουλειών μπορούμε να τα βελτιώσουμε όλα αυτά. Αναφερόμενοι στην ενέργεια πράγματι είναι εφικτό με την ευφυή τεχνολογία και τον τρόπο μέτρησης κατανάλωσης να μειώσουμε την κατανάλωση. Και η βιωσιμότητα μπορεί να επιτευχθεί μέσω της κατάλληλης τεχνολογίας να μπορέσουμε όλα αυτά να τα προωθήσουμε. Και αυτό με ενδιαφέρει πραγματικά. Όχι μόνο για... Δεν είναι θέμα μόνο ευμαρίας, αλλά είναι και θέμα ασφαλείας στην κινητικότητα, ε, βιωσιμότητα, είναι θέματα υγείας, είναι ενέργεια, νερό, τι θέλετε. Πρωτοβουλίε και σε αυτόν τον τομέα χρειάζονται. Εάν με υποστηρίξετε, θα πρέπει να συζητήσουμε, πιστεύω, στο νέο μας πρόγραμμα, το πρόγραμμα 8 για την έρευνα, ποιες είναι οι προτεραιότητες. Ξέρω ότι ίσως είναι παρακινδυνευμένα αυτά τα σχόλια που κάνω, όμως Μέχρι τώρα υποστηρίζω περισσότερο να παίρνουμε δύο μόνο θέματα που είναι πολύ σημαντικά και εκεί να ηγηθούμε, εκεί που έχουμε την αριστεία και να μην ε, διασπείρουμε τις προσπάθειές μας. Ποτέ δεν θα βρεις όλους τους φίλους με, από το μέρος σου αν δεν έχεις το θάρρος. Μπορεί να τους πεις η ιδέα αυτή είναι καλή αλλά όχι για αυτή τη στιγμή και θα πρέπει να προχωρήσουμε σε κάποιους τομείς κάνα δύο βήματα πρώτα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κυρία Υποψήφια Επίτροπες, στις γραπτές σας απαντήσεις και το είπατε και στην αρχή της ομιλίας σας, Είπατε ότι θέλετε να γεφυρώσετε το ψηφιακό χάσμα, ιδίω σε ό,τι αφορά τι πιο τροτέ ομάδε του πληθυσμού. Θα ήθελα να ξέρω ποια είναι η πρόθεσή σα λοιπόν για τα νοικοκυριά που έχουν χαμηλό εισόδημα, για του ηλικιωμένου, του άνεργου και του νέου, <clears throat> ώστε να μην βρεθούν σε κατάσταση κοινωνική μειονεξία όταν εμείς δημιουργούμε μια κοινωνία που βασίζεται στην ψηφιακή πληροφορία. Μια μελέτη η οποία έγινε από το Ιρλανδικό Πανεπιστήμιο του Κόρκ με τη βοήθεια τη Eurostat λέει ότι ίσως μπορεί να προκύψουν νέε κοινωνικέ ανισότητες γιατί ορισμένε κοινωνικές ομάδες δεν είναι σε θέση να χρησιμοποιήσουν υπολογιστές και ε, τεχνολογίες πληροφορίες. Ποια είναι η άποψή σας κυρία Κρούζ. <clears throat> Είμαι ικανοποιημένη με το ερώτημά σας. Ένα από αυτά τα θέματα που πρέπει να αντιμετωπίσουμε είναι καταρχήν το γεγονός ότι δεν ζούμε πια με τα δίκτυα και τα ψηφιακά μέσα, αλλά μέσα στα δίκτυα και μέσα στα ψηφιακά μέσα. Δεν είναι αυτό στο οποίο είχαμε συνηθίσει στο παρελθόν, όπου κάποιοι από εμά ήταν σε θέση ή θέλαν να λειτουργήσουν με αυτά τα μέσα. Αυτό είναι τώρα κομμάτι της ζωής μας, τούτου λεχθέντος. Και αυτό φυσικά είναι μία από τις προκλήσεις αυτού του χαρτοφυλακίου. <clears throat> Υπάρχουν ομάδες οι οποίες είναι κοινωνικά ορατές και εντοπίσιμες και μπορεί να είναι και θέμα ηλικίας φυσικά που δημιουργεί ομάδες μειονεκτικές. Είναι κρίμα λοιπόν να χάσουμε ολόκληρες γενιές επειδή τα πράγματα προχωρούν τόσο γρήγορα. Πρέπει να βοηθήσουμε λοιπόν τους πιο ηλικιωμένου και να τους βοηθήσουμε να μην φοβούνται. Γιατί μπορεί να είναι μεγάλη πίεση πάνω τους από την ψηφιακή αυτή κοινωνία. Και επίσης στα κράτη-μέλη θα πρέπει να υπάρξει συνεισφορά αν εξασφαλιστεί η ύπαρξη ευρυζωνικών συνδέσεων παντού. Δεν μπορεί κανείς να ισχυριστεί ότι δεν λαμβάνει υπόψη τις ανάγκες αυτών των ομάδων και των στρωμάτων του πληθυσμού. Πρέπει να προχωρήσουμε και με εκπαιδευτικά μέτρα και είμαι σίγουροι ότι κάποιοι από εσά έχουν διαβάσει το άρθρο αυτό στους New York Times για την Δανία, για την υγειονομική περίθαλψη. Μπορεί να είναι πολύ σημαντική λοιπόν η χρήση των ψηφιακών τεχνολογιών για τα άτομα τα ηλικιωμένα. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό λοιπόν να δώσουμε τέτοιες ε, ευκαιρίες. Ας είμαστε λοιπόν <clears throat> επάγρυπνοι για να βοηθήσουμε αυτούς οι οποίοι δεν ξέρουν ακόμα πόσο σημαντικά είναι τα ψηφιακά μέσα στην εποχή μας. Συμπληρωματικό ερώτημα παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ για την απάντησή σας. Έχω άλλη μία ερώτηση που εφήγει από κάποιους από κάποιους συμπατριώτες σας από την πολιτική μου ομάδα, από τον κύριο Ντένις Δε και το ερώτημα αφορά τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Μόνο 10% των μικρομεσαίων επιχειρήσεων συμμετέχουν στα ε, ψηφιακά δίκτυα υψηλής ταχύτητας. Πώς μπορείτε να προστατεύσετε πολύ καινοτόμε ε, μικρέ, μικρομεσαίε επιχειρήσει που καταβροχθίζονται από μεγαλύτερε. Απάντηση. Ένα βασικό μου στόχο, κάτι αγαπημένο σαν θέμα. Όταν ήμουν υπεύθυνη για την πολιτική ανταγωνισμού και για τι κρατικέ ενισχύσει εστιάστηκα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι 99% των επιχειρήσεων στην Ευρώπη. Αν θέλουμε να αυξήσουμε τις θέσεις απασχόλησης και να αναπτυχθεί η οικονομία, αυτές είναι που δημιουργούν τις θέσεις εργασίας και όχι κυβερνήσεις και τίποτα άλλο. Τούτου λεχθέντος. Πρέπει να τις πάρουμε στα σοβαρά. Με τα μέτρα κρατικών ενισχύσεων δίνουμε κάποιο ανατολισμό στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Αυτό μπορεί να συνδεθεί και με αυτό που συζητάμε. Και να υπάρχει η δυνατότητα κρατική ενίσχυσης για ευρυζωνικά δίκτυα. Εγώ θα ήθελα να εστιαστώ όχι μόνο στο να τις παροτρύνουμε να χρησιμοποιήσουμε αυτά που υπάρχουν, αλλά να προωθήσουμε την καινοτομία και την έρευνα σε αυτούς τους τομείς Θέλουμε όπως με την Apple να μπουν στα γκαράζ, να θέλετε, στα δωμάτια του και τα αγόρια και τα κορίτσια και να, επι... να δημιουργούν καινοτομίε, να εφευρίσκουν προϊόντα κλπ. Θέλουμε λοιπόν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και αυτές να συμμετάσχουν και να χρησιμοποιήσουν τις νέες δυνατότητες που υπάρχουν και να προωθήσουμε την καινοτομία και την έρευνα. Και πολύ συχνά είναι θέμα να τους πρόξουμε να δραστηριοποιηθούν. Υπάρχουν οι δυνατότητες. Ο Κυρία Κρούς, θα σας θέσω το, την ερώτηση στα ελλανδικά στην τρική σας γλώσσα. Καταρχάς, να σας πω ότι σας ε, συγχαίρω για τον διορισμό την υποψηφιότητά σας για τη θέση αυτά. Θα ήθελα να σας ρωτήσω για την εσωτερική αγορά. Η εσωτερική αγορά δεν είναι σωστή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν λαμβάνονται τις ευκαιρίες όλες οι εταιρείε. Η Γερμανία προστατεύει τις γερμανικές επιχειρήσεις, η Γαλλία τις γαλλικές επιχειρήσεις και σε κάποιες περιπτώσεις οι Ολλανδικές επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν προβλήματα. Προβλήματα, για παράδειγμα, αντιμετωπίζουν επιχειρήσεις ε, Ολλανδικές του κλάδου τηλεπικοινωνιών. Τι θα κάνετε λοιπόν, σας ερωτώ, για να δημιουργήσετε ίσους όρους ανταγωνισμού για το τομέα των τηλεπικοινωνιών. Γιατί το κόμμα για την ελευθερία θεωρεί ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχουν ίσοι όροι ανταγωνισμού και σας ερωτώ λοιπόν τι σκοπεύετε να κάνετε για να το διαβαλήσετε αυτό. Κύριε Πρόεδρε, ο αξιότιμος βουλευτής ε, υποδεικνύει για μία φορά ακόμα πόσο σημαντικό είναι να μην μιλάμε μόνο τυπικά και στα χαρτιά για μια νέα αγορά χωρίς σύνορα, αλλά κάτι τέτοιο να ισχύει και στην πράξη, να λειτουργεί στην πράξη. Συμφωνούμε απόλυτα ότι ασφαλώς δεν έχουν πραγματοποιηθεί, δεν έχουν υλοποιηθεί όλα όσα θα έπρεπε να έχουν υλοποιηθεί και θα είμαι τελευταία που θα πει Μάλλον μετά είμαι καν η τελευταία που θα πει ότι έχουμε ακόμα πολλά να κάνουμε. Αλλά είμαι λίγο λιγότερο αρνητική από είστε εσεί. Δεν ε, μιλώ για τον τομέα των τηλεπικοινωνιών. Μιλώ για το σύνολο τη αγορά. Αυτό που είδαμε στο τρέχον χαρτοφυλάκιό μου είναι ότι από καιρό ει καιρό και σίγουρα όταν υπάρχει δύσκολη οικονομική κατάσταση υπάρχουν τάσεις προστατευτισμού, αλλά ως τώρα πρέπει να σας ε, πω, όταν μας γνωστοποιείτε κάτι τέτοιο, αναλαμβάνουμε δράση και οι αντιδράσεις είναι θετικές. Και ξέρουμε εντωμεταξύ ότι από πλευρά Βρυξελών, από πλευρά Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θα αναλυφθεί δράση και ότι δεν είναι δυνατόν να λειτουργήσει κανεί σε αντίθεση με του κανόνε μα. Τώρα, συγκεκριμένα για τι ε, επιχειρήσει τηλεπικοινωνία, γιατί σε αυτέ εστιάσατε πιο συγκεκριμένα και δικαίω. Όντω, η απελευθέρωση των επιχειρήσεων των υπηρεσιών αυτών ήταν μια φανταστική εξέλιξη, αλλά σε κάποιες χώρες δεν ε, τη χάνει τη μεταχείριση τη οποία ε, θέλαμε εμεί στην ενιαία αγορά προκειμένου να ισχύουν ίσοι κανόνε ανταγωνισμού. Τι θα κάνω, ρωτάτε. Θα είμαι πάρα πολύ. Θα επαγρυπνώ για να δω τι γίνεται και τι συμβαίνει στην πραγματικότητα. Δεν θα πιστεύω τον καθένα που θα βγαίνει και θα λέει ότι α, υπάρχει δίκαιος ανταγωνισμός και θα αντιδράσω με σαφήνεια για να δω τι θα μπορέσουμε να κάνουμε. Να, θα μιλήσω με, τους, με τις επιχειρήσεις, με τις χώρες και θα πρέπει να τηρηθούν οι κανόνες. Πολύ απλά δράσιμη η απάντησή μου. Έχετε άλλη ερώτηση? Όχι, νομίζω ότι ήταν πολύ σαφή η απάντηση, δεν έχω κάποια άλλη ερώτηση. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε κύριος σας ευχαριστώ, Πρόεδρε, αξιότιμη κυρία Επίτροπε. Χαίρομαι που σήμερα εδώ στην Ακρόαση διευκρινίστηκαν κάποια θέματα. Θα ήθελα να σας ρωτήσω ποια είναι η διαφορά μεταξύ της αξιολόγησης, της περιαγωγής μεταξύ της Επιτρόπου Ανταγωνισμού και της Επιτρόπου για την ψηφιακή ατζέντα, για το ψηφιακό πρόγραμμα δράσης. Θα ήθελα να αναφέρω το θέμα της περιαγωγής δεδομένων. Διαπιστώσαμε ότι Υπάρχουν, ε, για παράδειγμα, σε χοντρικό εμπόριο 1 ευρώ, ε, τιμολογία 1 ευρώ την ώρα και στο, στη χώρα μου ισχύει, στη χώρα μου ισχύει το 1 λεπτό και κοιτώντας τι γίνεται στο Βέλγιο, βγαίνοντας δηλαδή από τη χώρα μου, πληρώνω 13 λεπτά για την ίδια υπηρεσία. Δηλαδή για την ίδια υπηρεσία να πληρώνω ή ένα λεπτό ή ένα ευρώ ή 13,9 ευρώ. Βλέπω λοιπόν ότι υπάρχει ένα τέτοιο όριο κατάχρησης. Οι πιο πολλές επιχειρήσεις τηρούν το όριο κατάχρησης του 0,25. Έχουμε τα 4 λεπτά. Πώς ε, θεωρείτε ότι αυτή η διαφορά μεταξύ της θέσης σας ως Επιτρόπου για τον ανταγωνισμό και για την ψηφιακή ατζέντα θα μπορέσει να α, συμψηφιστεί. Απάντηση. Ε, ε, ελπίζω να είμαι συνεπής. Αν με υποστηρίξετε δεν θα υπάρχει μεγάλη διαφορά. Θα ήταν παράξενο διαφορετικά. Κύριε Πρόεδρε, ξέρω ότι απαντώ σε ένα επιφανέστατο μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για θέματα ε, περιαγωγής. Ξέρω ότι ξέρετε τα πάντα για αυτό το θέμα. Κατά παρελθόν μου είχατε δώσει πληροφορίες που ε, μου έδειξαν πληροφορίες ότι δεν έχουμε φτάσει εκεί που θέλαμε. Αυτό που πετύχαμε, αυτό κάθε αυτό είναι πολύ καλό. Συγχαρητήρια στην κυρία Ρέντινγκ, συγχαρητήρια στο Κοινοβούλιο. Ήταν καλή συνεργασία, πραγματική συνεργασία και είμαι σίγουρη ότι έχοντας κάνει αυτά τα δύο βήματα στις δύο αποφάσεις του 2007 και του 2009 καταφέραμε πολλά. Τώρα φάγαμε το γάιδρο μένει ουρά. Αναφερθήκατε στο θέμα για τα δεδομένα και λοιπά που σας ανησυχεί. Πρέπει να συνεχίσουμε. Ιδεώδεις λύσεις θα ήταν ευρωπαϊκή αγορά περιαγωγής χωρίς σύνορα. Δεν είμαι σίγουρη αν αρκούν πέντε χρόνια για κάτι τέτοιο. Ούτε ξέρω αν δεν φτάνουν τα πέντε χρόνια. Αλλά είναι πρόκληση ο στόχος για τον καταναλωτή στην εταιρική αγορά τηλεπικοινωνιών. Η διέλευση εσωτερικών σύνορων δεν θα έπρεπε να έχει κάποιο αποτέλεσμα ή ελάχιστη διαφορά όσον αφορά τις παρεχόμενες υπηρεσίες και την τιμή αυτών. Πρέπει να περιμένουμε τα αποτελέσματα της μελέτης, να αναλύσουμε τα αποτελέσματα, να δούμε τι γίνεται και μετά το Μάρτιο θα μπορέσουμε να επικοινωνήσουμε, αν βέβαια κατέχω αυτή τη θέση, αν έχω επικυρωθεί στη θέση της ε, Επιτρόπου ερώτηση ο Σας ευχαριστώ. Αυτό σημαίνει δηλαδή θα προτείνετε ενδεχομένω ε, κανονισμό, τρίτο κανονισμό για, το, για την περιαγωγή, για το roaming. Οι ειδικέ σα αποφάσει που αφορούν το πακέτο τηλεπικοινωνιών μας δείχνουν ότι με τις εθνικές ρυθμιστικές αρχές δημιουργείται νέος χώρος όχι μόνο για σας είναι καινούργια τα πράγματα με το πρόγραμμα της Λισαβόνα που έχετε αυξημένες εξουσίες τώρα, αλλά όσον αφορά αυτό το τομέα και για αυτές τις αρχές με στενή συνεργασία που είναι μεγάλη πρόκληση, συνεργασία με εθνικές ρυθμιστικές αρχές και με το Κοινοβούλιο θα πρέπει να κινηθούμε, να περιμένουμε την διάμεση έκθεση το καλοκαίρι και με τελική έκθεση που θα έχουμε στα χέρια μας μετά από ένα χρόνο, θα έχουμε ξεκάθαρα συμπεράσματα, ελπίζω. Ο κανονισμός για την περιαγωγή δεν θα πρέπει να είναι ο δικός μου στόχος. Για πάντα. Η αγορά θα πρέπει να τα ρυθμίζει και όχι ε, εκ των άνω. Αλλά θα πρέπει να το αξίζει η αγορά, να μπορεί να αυτορυθμίζεται η αγορά της περιαγωγής. Κυρία Ευχαριστώ πολύ. Βλέπω ότι έχετε ένα μεγάλο ερωτηματικό στο ταγέ σας. Δεν ξέρω πώς πρέπει να το ερμηνεύσω. Νομίζω ότι απλώς συμβολίζει ότι κάποιοι θέτουν ερωτήσεις και εσείς δίνετε απαντήσεις. Και εγώ θέλω να σταθώ στο θέμα της ουδετερότητας του διαδικτύου. Είναι πολύ μεγάλη σημασία για μένα. Η Κομισιόν έχει, επί τη βάση μιας πρωτοβουλίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της Κατρίν Τρότμαν συγκεκριμένα, έχει ξεκινήσει ένα έλεγχο, μια έρευνα της κατάστασης αυτής και δεν ξέρουμε ακόμα ποια θα είναι τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας. Αλλά ξέρω ότι η Κομισιόν έχει ήδη προετοιμάσει ένα έγγραφο προβληματισμού σε σχέση με την ε, ουδετερότητα στο διαδίκτυο και φαίνεται ότι είναι ένα κάπως συγκεχημένο ε, έγγραφο. Μπορείτε να μας πείτε κάτι για όλα αυτά, κύριε Κρούς. Το πιο εύκολο κομμάτι να απαντήσω, κύριε Πρόεδρε, είναι η καρφίτσα μου. Πράγματι, είναι διαλαγμένη. Διάλεξα επίτηδε. Όχι ότι δεν κάνω ό,τι μπορώ για να απαντήσω τα ερωτήματά σα. Για αυτήν έχω, διότι δεν είμαι σίγουρη. Το ερωτηματικό φορά το αποτέλεσμα τη ακρόαση. Αυτό είχα υπόψη μου όταν έβαλα αυτή την καρφίτσα. Τούτου λεχθέντος. Αυτή η ενδιάμεση έκθεση, περί τίνος πρόκειται. Δεν ξέρω ποια θα είναι τα τελικά πορίσματα, να το πω έτσι. Εγώ θα ακολουθήσω τη γραμμή μου. Πρέπει να ε, ε, ε, ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα της αγοράς και διαφάνεια. Θέλουμε ανοιχτό και ουδέτερο δίκτυο. Αλλιώς χάνονται δυνατότητες. Το ανέφερα και προηγουμένως, όταν απαντούσε την κυρία Λαμπέρ. Και αυτό θα πρέπει να ληφθεί υπόψη. Ουδετερότητα του δικτύου είναι το βασικό ζήτημα. Δεν πρέπει να ακολουθήσουμε άλλο δρόμο από αυτόν. Ο Συμπληρωματικό ερώτημα, κύριε Όλσκοκ. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ για την απάντησή σας κυρία Κρούζ. Αλλά ίσως η σύγχυση για το έγγραφο αυτό μπορεί να προκύπτει από το γεγονός ότι υπάρχουν διαφορετικοί ορισμοί για την έννοια της ουδετερότητας στο διαδίκτυο. Τι σημαίνει για σας η ουδετερότητα αυτή, ποιος είναι ο ορισμός η ουδετερότητα στο διαδίκτυο. Για μένα η ουδετερότητα του δικτύου Και καταλαβαίνω ότι λέτε, ότι επικρατεί σύγχυση όσον αφορά αυτό. Δεν είναι ξεκάθαρος ορισμός. Λοιπόν, για μένα, το σημαντικό είναι κατά πόσο η πρόσβαση στο διαδίκτυο, ή μάλλον οι παρέχοντες υπηρεσίες διαδικτύου, μπορούν να ελέγχουν ή να περιορίζουν τους χρήστες, την πρόσβαση των χρηστών σε κάποιο περιεχόμενο. Όταν αυτό γίνεται λόγω εμπορικών κινήτρων, αυτό είναι απαράδεκτο. Μόνο αν είναι θέμα ασφάλειας. Ή αν επιθύματα μηνύματα, spam, αλλά τέλος πάντων για άλλους λόγους και μη εμπορικούς. Γιατί διαφορετικά αν για άλλους σκοπούς γίνεται διήθηση των, του, της πρόσβασης, τότε είναι απαράδεκτο. Thank you very much. Um, Ο συνάδελφος ευχαριστώ πολύ και ένα από τα πιο σημαντικά και δύσκολα θέματα για τα επόμενα χρόνια είναι πώς ε, θα γεφυρώσουμε το ψηφιακό χάσμα για το πώς θα προάγουμε την Ευρώπη ως ηγετική περιοχή του κόσμου σε ό,τι αφορά τις τεχνολογίες πληροφοριών κάθε είδους. Πώς πρόκειται λοιπόν να προχωρήσετε σε ό,τι αφορά το ψηφιακό χάσμα προφανώς, για, προφανώς προκειμένου να διασφαλίσετε ότι το ψηφιακό φάσμα θα δώσει ευκαιρία σε όλες τις διαφορετικές υπηρεσίες στην Ευρώπη. Απάντηση. Κάποιες φορές, κύριε Πρόεδρε, Βλέπω ότι έχω πολλά θετικά στοιχεία και έχω λοιπόν μια μεγάλη ευκαιρία σε ό,τι αφορά το ψηφιακό χάσμα. Η ευκαιρία αυτή έγκυται στην αλλαγή συστήματος. Αυτό αποτελεί μια μεγάλη ευκαιρία. Η αλλαγή, η μετάβαση από την λογική στην ψηφιακή τηλεόραση. Αυτό θα δώσει στις εταιρείε ε, την δυνατότητα να αναπτύξουν και να προωθήσουν τις υπηρεσίες τους. Θα πρέπει όντως να χρησιμοποιηθεί στη συγκεκριμένη περίσταση η εσωτερική αγορά και να γίνει όσο το δυνατόν μεγαλύτερη εναρμόνιση γίνεται. Γιατί αν τα κράτη-μέλη δράσουν με διαφορετικό τρόπο θα χάσουμε πολλές πτυχές. Άρα η αποτελεσματική και αποδοτική χρήση του φάσματος συμβάλλει στην ε, υλοποίηση της πολιτικής μας και θα μπορούσε να παρέχει μεγαλύτερη ποιότητα πολλές περισσότερες ευκαιρίες και δυνατότητες και θα έπρεπε να, να αναφέρουμε δύο διαφορετικά στοιχεία. Επιτρέψτε μου να το αναφέρω. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζητάει από τα κράτη-μέλη να ολοκληρώσουν ε, τις διαδικασίες για το κλείσιμο της αναλογικής τηλεοράσης και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ορίσει και σχετικό χρονοδιάγραμμα μέχρι το 2012 και κατά δεύτερον θα πρέπει να υπάρχει συντονισμένη δράση από τις εθνικές αρχές για να ανοίξει το φάσμα για ανταγωνιστικές νέες υπηρεσίες. Και πρόκειται να διαθέσουμε ε, εναρμονισμένους όρους για τα κράτη-μέλη που σκοπεύουν να ανοίξουν το φάσμα των 800 MHz για τις ε, υπηρεσίες αυτές πέρσι τον Οκτώβριο. Έγινε μια συντονισμένη δράση από τις εθνικές αρχές για να ανοίξει το φάσμα σε καινοτομικές και ανταγωνιστικές νέες υπηρεσίες και εμείς προωθήσαμε την δράση αυτή. Άρα στο σύνολο πρέπει να παρατηρήσουμε ότι υπάρχουν ε, πολλές ε, προκλήσεις. Ε, ερώτηση, συμπληρωματική ερώτηση από τον κύριο Χόκμαρκ. Ευχαριστώ πολύ. Αυτό είναι θετικό, αλλά θα ήθελα και να υπογραμμίσω το ερώτημα του τι θα κάνετε με τη διαδικασία εκχώρησης. Πώς θα διασφαλίσετε ότι θα αντιμετωπίσετε τις συγκρούσεις συμφερόντων σε ό,τι αφορά τα παραδοσιακά συμφέροντα, αλλά και τις ε, νέες κινητομικές ευκαιρίες. Νομίζω ότι αυτό θα είναι πολύ σημαντικό θέμα. Και θα είναι και καθοριστικό για να επιτευχθεί μια ενιαία ψηφιακή αγορά στην Ευρώπη. Αν θέλουμε στο μέλλον να αποφύγουμε τα εθνικά συστήματα περιαγωγή, θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε αυτό το ψηφιακό πλεονέκτημα. Απάντηση. Θα ήθελα να τονίσω τρία στοιχεία. Καταρχάς, ε, η Σύνοδος για το φάσμα που θα, που θα διοργανωθεί από την, ε, το Κοινοβούλιο, την Επιτροπή και το Συμβούλιο μετά από πρωτοβουλία του Κοινοβουλίου και είναι εξαιρετικά χρήσιμη πρωτοβουλία. Κατά δεύτερον, μετά από την σύνοδο αυτή θα πρέπει να προετοιμαστούν τα σχετικά συμπεράσματα και ένα πρόγραμμα πολιτικής για το ραδιοφάσμα επί πολιετούς βάσης και μετά να βοηθηθούν τα κράτη-μέλη να εντοπίσουν τις διαφορές. Αλλά επίσης να έχουμε υπόψη μας ότι με θέματα ουδετερότητας ε, του δικτύου οι παλαιοί φορεί δεν θα τύχουν μετάχειρίσεις μεταχείριση σε σχέση με τους καινούριου. αλλά το ίδιο ισχύει και αντιστρόφως. Άρα θα υπάρχει μια διαδικασία εποπτείας και σε τελική ανάλυση τα συμπεράσματα θα πρέπει να είναι θετικά. Αν δεν είναι θετικά θα πρέπει να υπάρξει διορθώση. Ευχαριστώ κυρία Τικάου έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Επίτροπε. Κυρία Επίτροπε, ελπίζω ότι το ερωτηματικό στο φόρεμά σας δείχνει ότι είσαστε ανοιχτοί στο διάλογο και ότι έτσι μπορούμε να βρούμε απάντηση σε πολλά ερωτήματα. Το δικό μου ερώτημα είναι το εξή. Οι αγορέ του διαδικτύου χρειάζονται μια αποτελεσματική διοικητική διαδικασία συνεργασίες. Και ξεκινώντας με τον Ιανουάριο του 2010 προβλέπει η αρμόδια οδηγία ότι όλοι οι πάροχοι υπηρεσιών θα πρέπει να έχουν πρόσβαση στις κατάλληλες πληροφορίες, να υπάρχει ένα συγκεκριμένο και μοναδικό σημείο πρόσβασης, το οποίο θα είναι ηλεκτρονικά προσβάσιμο. Αυτός ο στόχος όμως δεν έχει επιτευχθεί ακόμα λόγω νομικών και τεχνικοδιοικητικών προβλημάτων. Υπάρχει ανάγκη ψηφιακών πιστοποιητικών για να λάβει κανεί μέρος σε ένα τέτοιο διαγωνισμό. Θα ήθελα να σας ρωτήσω ποια είναι η κατάσταση για το πρόγραμμα αυτό που έπρεπε να ξεκινήσει το 2010 και τι θα κάνετε για να εξασφαλίσετε την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας μέσα από την ανάπτυξη της κοινωνίας των πληροφοριών και μιλώ περισσότερο για την ε, ηλεκτρονική διακυβέρνηση, του ηλεκτρονικούς λογαριασμούς, τις ευρωζωνικές υπηρεσίες κτλ. Κυρία Κρούζ, έχετε το λόγο. Πράγματι, το χρονοδιάγραμμα δεν τηρήθηκε πλήρως όπως είχαμε υποσχεθεί. Αυτός όμως δεν είναι ε, λόγος να αλλάξουμε γραμμή πλεύσης. Έχετε εξηγήσει κι εσείς τι εμπόδισε την εφαρμογή αυτού του χρονοδιαγράμματος, αλλά είναι, εν η απόλυτη προτεραιότητα για τους παρόχους υπηρεσίες να ξέρουν ότι αν αυτοί τηρούν τους κανόνες και οι συνεργάτες τους και οι, συνομιλητέ τους κατά κάποιο τρόπο και αυτοί τηρούν τους κανόνες. Εγώ θα παρακολουθήσω αυτό το θέμα πάρα πολύ προσεκτικά και θα προωθήσω αυτά τα οποία είναι απαραίτητα και αν αυτό δεν είναι δική μας αρμοδιότητα θα πρέπει να υπάρξει και συζήτηση με τους εθνικούς ρυθμιστικούς φορείς και με εσάς ως Κοινοβούλιο εξάλλου. Ευχαριστώ κύριε Τικάου και πάλι. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Από ό,τι καταλαβαίνω λοιπόν το σχέδιο ε 2010 θα συνεχίσει με περαιτέρω φιλόδοξου στόχου. Απλώ θέλω να σας υπενθυμίσω επίση το γεγονός ότι η ανάπτυξη μιας <clears throat> υποδομής επικοινωνιών και η προσβασιμότητα των συστημάτων πληροφόρηση και επικοινωνιών που να εγγυάται την ασφάλεια των επικοινωνιών και να σέβεται τα δικαιώματα των χρηστών, όλα αυτά είναι απαραίτητα και απαράγραπτα για την κοινωνία των, των πληροφοριών. Πέρσι 40% των Ευρωπαίων δεν χρησιμοποίησαν το ίντερνετ και 46% των οικοκυριών δεν είχαν πρόσβαση στο ίντερνετ. Τι μέτρα προβλέπετε να λάβετε για να μπορέσετε να επιτυχείτε το στόχο της κάλυψης 100% για το ευζωνικό ίντερνετ ακόμα και σε απομονωμένες περιοχές. Και τι θα κάνετε για τα άτομα με αναπηρίες. Λοιπόν, τέσσερις ερωτήσεις. Κύριε Πρόεδρε, να απαντήσω στο πρώτο ερώτημα. Ναι, ή 2010 θα προχωρήσουμε στην πορεία που έχουμε καθορίσει. Γιατί δεν χρησιμοποιούν όλοι τις δυνατότητες που παρέχονται. Και δεν μιλώ για τις περιοχές που δεν καλύπτονται 100% αλλά αυτές που καλύπτονται. Υπάρχουν υπηρεσίες, αλλά δεν χρησιμοποιούνται. Ένα-δύο πράγματα που θα μπορούσαν να κάνουν τη διαφορά είναι η εμπιστοσύνη και η ασφάλεια. Και ήταν ενδιαφέρον που ανακάλυψα αναφερόμενοι στις οικονομικές δραστηριότητες ή δραστηριότητες πραγματικά πρέπει να υπάρχει ασφάλεια να είσαι σίγουρος ότι δεν γίνεται κατάχρηση ιδιωτικών δεδομένων κλπ. Αυτό θα πρέπει να τονιστεί, να το προσέξουμε. Διότι αν υπάρχει υπάρχει καχυποψία από πολλούς ανθρώπους και χρειάζεται εκπαίδευση, δεν θέλω να χρησιμοποιώ αυτόν τον όρο, να ενημερώσουμε τον κόσμο περί πρόκειται και καμιά φορά χρειάζεται πολύ μεγαλύτερη προσοχή από τη δική μας πλευρά και από την πλευρά των κρατών μελών. Καμιά φορά λείπει ευαισθητοποίηση. 100% ευρυζωνική κάλυψη. Θα κάνω ό,τι μπορώ να συναθρήσω τα εμπλεκόμενα μέρη να ετοιμάσουμε σχέδια. Δεν είναι πάντα στην ύπεθρο, δεν υπάρχει δυνατότητα να ακολουθηθεί συγκεκριμένη λύση. Με κρατικές ενισχύσεις ίσως μπορεί να καλυφθεί αυτό το πρόβλημα, να καλυφθεί, να υπάρξει 100% κάλυψη. Τα άτομα με αναπηρία, αυτό είναι στον κατάλογο κάθε προσπαθίας Ευρωπαϊκής. Αγαπητοί συνάδελφοι και κυρία Κρούς, πρέπει οπωσδήποτε να τηρήσουμε τον χρόνο. Δεν θέλουμε να μείνουν οι τελευταίοι χωρίς δυνατότητα να θέσουν ερωτήματα. Σας παρακαλώ να είσαστε προσεκτικοί για τον ε, χρόνο σας. Ο κύριος Κανσιάν έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε υποψήφια. Ε, Κυρία Υποψήφια Επίτροπε, έχετε πολύ σημαντικό χαρτοφυλάκι, όλα πολύ ευαίσθητο, βιώσιμη ανάπτυξη. Καλύπτεται εδώ, θα πρέπει να εγγυηθείτε την ασφάλεια και τι παραβιάσεις ή οδήποτε είδου και παρατυπίες, παραποίηση θα πρέπει να αποφύγετε και θα πρέπει να προστατεύονται τα ιδιωτικά στοιχεία, η ιδιωτική ζωή. Θέλω να περιστώ εδώ στα δικαιώματα του δημιουργού. Η ψηφιοποίηση των λογοτεχνικών έργων και των ηλεκτρονικών βιβλίων και των διαφόρων δοκιμίων των πανεπιστημιακών είναι πολύ προχωρημένα, όμω δεν προστατεύονται ε, παρκώς το πνευματικό δικαίωμα. Υπάρχει ανεπάρκεια όσον αφορά την οδηγία 29 του 2001 να καλύψει όλο τον τομέα. Και τα κράτη-μέλη βρίσκονται σε αδύναμη θέση όσον αφορά την αγορά έναντι άλλων αγορών όπως είναι η Αμερικανική αγορά. Υπάρχουν υποχρεωτικές εξαιρέσεις όσον αφορά τα δικαιώματα του δημιουργού. Πώς προτίθεστε κυρία Επίτροπε, υποψήφια Επίτροπε, να προσαρμόσει την κοινοτική νομοθεσία και να μπορεί να προσαρμοστεί στην τεχνολογική πρόοδο και αυτές οι γενικές εξαιρέσεις ε, μπορεί, μπορεί τελικά να ρυθμιστούν ούτως ώστε να υπάρχει καλύτερη κάλυψη ε, όσον αφορά τα πνευματικά δικαιώματα και αφορά το θέμα αυτό τη διδασκαλία και την ε, τεχνική και την κατάρτιση. Απάντηση. Ένα από τα ευαίσθητα κομμάτια είναι τα πνευματικά δικαιώματα της, στην πολιτική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Μιλώντας για πειρατεία, είναι ένας κύκλος. Όσο υπάρχουν κατακαιρματισμένοι κανόνε, σε εθνικό επίπεδο διαφορετικοί κανόνε για πνευματική ιδιοκτησία, είναι δύσκολα τα πράγματα. Είναι πολύ δύσκολο να έχει κανεί μια πρωτοβουλία ευρωπαϊκή κατά τη πειρατεία. Αυτό δεν είναι το μόνο ζήτημα. Συμφωνούμε όλοι ότι εκείνοι που δημιουργούν μια υπηρεσία, ένα προϊόν, αξίζουν να πληρωθούν. Τούτου λεχθέντος, αν δεν καταφέρουμε να χρησιμοποιήσουμε την πρόκληση της προσέγγισης ενιαίας αγοράς, τότε θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να βρούμε έναν τρόπο με τον οποίο να κάνουμε αυτό που πρέπει. Και προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα, είναι σημαντικό αυτό για την οικονομία, για τον πολιτισμό και οι δημιουργοί το αξίζουν. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα εξακολουθεί να παρακολουθεί τις πρωτοβουλίες των κρατών μελών, θα προωθήσουμε τις νομικές επιλογές προσφέροντας ευρία επιλογή για τους καταναλωτές και θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας από αυτό που κατάλαβα, αυτό που είπε και ο κύριος Μισελ Μπαρνιέ, είναι ότι και αυτός ενδιαφέρεται να βρει μια λύση. Θα προσπαθήσουμε να συνεργαστούμε και να κάνουμε ένα βήμα μπροστά. Αυτό που φοβούμε, και αυτό είναι το τελευταίο που έχω να πω, είναι ότι οι άλλοι μας περνούν και η Ευρώπη επειδή δεν λύνει αυτό το πρόβλημα, μένει πίσω. Τελευταία. Κύριο Κάνσιαν, ανάλλη μια ερώτηση. Ε, τρία, δευτερόλεπτα. Με ικανοποιεί απάντηση, αλλά προσοχή στο χρονοδιάγραμμα, διότι είναι σημαντικός ο χρονισμός όσον αφορά το ευαίσθητο αυτό θέμα και θα ήθελα απλώς να σας ζητήσω να είστε διαθέσιμοι να ευνοήσετε τις τεχνολογίες κυρίως όσον αφορά την πρόσβαση στους, να μπορούν οι, άνθρωποι που έχουν πρόβλημα όρασης και οι τυφλοί να έχουν πρόσβαση σε λογοτεχνικά έργα. Απάντηση. Με τα χαράς να έχω την ευκαιρία να κάνω κάτι τέτοιο, σας διαβεβαιώνω. Κυρία Ρόλο, ευχαριστώ. Στη γραπτή σας απάντηση, η κυρία Χόλ, αναφέρεται ότι οι τεχνολογίες πληροφοριών είναι σημαντικές και για την αντιμετώπιση της αλλαγής του κλίματος και σε ό,τι αφορά τους ηλικιωμένους. Υπάρχουν πολλά προγράμματα τα οποία μπορεί να περιορίσουν την κατανάλωση ενέργειας, όπως για παράδειγμα στα κτίρια, στις μεταφορές, στις μεταφορές και στην, ε, στις προμήθειες. Τι πιστεύετε ότι μπορείτε να κάνετε προκειμένου οι τεχνολογίες αυτές να επισέλθουν και να προσθεθούν στην καθημερινή χρήση απάντηση. Το θέμα είναι οι επικοινωνίες και η επικοινωνία με τον κόσμο. Έχω σε κάποιες περιπτώσεις την εντύπωση ότι αν δεν χρησιμοποιήσουμε, δεν αξιοποιήσουμε την ευκαιρία για να εμπλέξουμε όλους τους φορείς στην διαδικασία αυτή, το αποτέλεσμα που επιτυγχάνουμε είναι πολύ χαμηλότερο. Υπάρχει πάρα πολύ δημιουργικότητα, πάρα πολύ ενδιαφέρον και θέληση για συμμετοχή. Ας ε, ενημερώσουμε λοιπόν τον κόσμο για το τι γίνεται και αυτό προσπάθησα και στο χαρτοφυλάκιο του ανταγωνισμού. Καταλαβαίνω ότι στο συγκεκριμένο χαρτοφυλάκιο του ψηφιακού προγράμματος ε, η πρόκληση θα είναι ακόμα πιο μεγάλη. Αλλά είμαι πρόθυμη να αντιμετωπίσω αυτή την, την πρόκληση. Κυρία Χολ, δεύτερη ερώτηση για την ε, τεχνολογία GPS. Είναι καλά εγκαθιδρυμένη, αλλά καμία τεχνολογία κατεπίγουσας βοήθειας στην Ευρώπη δεν μπορεί να συνδράμει πολίτες που βρίσκονται σε ανάγκη με την τεχνολογία αυτή. Έχετε κάποιο σχέδιο για να διασφαλίσετε ότι όλη η φυστάμενη τεχνολογία θα επιτεθεί στην υπηρεσία 112 για την διάσωση ζώων. Καταρχάς, ε, καταρχάς να κάνουμε το θετικό απολογισμό. Όλα τα κράτη-μέλη πλέον συμμετέχουν στην διαδικασία αυτή και έχουμε ορίσει και σχετική ημερομηνία. Θα πρέπει να ενημερώσουμε και πάλι το λοιπόν θέμα ενημέρωση στον κόσμο, αλλά στην τελική ανάλυση εξαρτάται από τα κράτη-μέλη να ερμηνεύσουν τη συμμετοχή τους σε αυτό το μεγάλο πρόγραμμα. Και θα πρέπει φυσικά να λάβουμε υπόψη ότι όντω σώζουμε ζωές, πολλές ζωές. Ευχαριστώ κύριε Σουκαλά. Να σας καλησπερίσω ερήτημος κυρία και να σας καλωσορίσω στο Ευρωκοινοβουλίο. Here ε, κάνοντας χρήση των τριών παρεμβάσεων των συναδέλφων που αναφέρθηκαν στην ουδετερότητα του δικτύου, θα ήθελα να συνοψίσω ρωτώντας σας τα ακόλουθα. Πρώτον, αν κατάλαβα καλά, είστε έτοιμοι να δεσμευτείτε για την προστασία του ουδέτερου χαρακτήρα του διαδικτύου. Θα ήθελα να μου πείτε ποιες είναι οι δράσεις που θα αναλάβετε για τη διασφάλιση αυτής της ουδετερότητας του ανοιχτού διαδικτύου δηλαδή για τους Ευρωπαίους πολίτες. Αναφερθήκατε επίσης στις παρεμβάσεις των ε, διαφόρων παρόχων στην παρεμπόδιση που θέτουν στην εφαρμογή του Voice over IP. Θα ήθελα να μας πείτε ποια, ποια μέτρα είστε διατεθειμένοι να λάβετε για αυτό το σημείο. Ευχαριστώ. Κυρία Κρούς, και πάλι από κοινού με τα κρατη και με τους εθνικούς ρυθμιστές θα εξαρτηθεί το σύστημα αυτό. Μιλώντας για ουδετερότητα, δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν μπορεί να γίνει το voice, το voice over IP και επίσης θα χρησιμοποιηθεί η ίδια υποδομή. Θα πρέπει λοιπόν να δράσουμε, να αναγκάσουμε τους ιδιοκτήτες και εδώ επανέρχομαι σε μια απάντηση που έδωσα και προηγουμένως ότι υπάρχει διαφορά μεταξύ της εμπορικής προσέγγισης για... αλλά θα πρέπει να πούμε ότι αυτό είναι παράνομο αντίκειται στους κανόνες. Είμαι απόλυτα πεπισμένη ότι από κοινού μπορούμε να το πετύχουμε αυτό, αλλά θα πρέπει να επιδείξουμε μία προθεμία και να λάβουμε δράση και να καταδείξουμε ότι είμαστε σοβαροί και ότι αυτή θα είναι η γραμμή που θα ακολουθήσουμε. Την έννοια, θεωρείτε ότι η ουδετερότητα του διαδικτύου θα πρέπει να αποτελεί επίσης δεσμευτική προϋπόθεση για τα νέα ευρωπαϊκά τηλεπικοινωνιακά δίκτυα ιδίω για αυτά που θα προκύψουν από την αξιοποίηση του digital dividend. In principle, I think Επί της αρχής νομίζω ότι θα πρέπει να τηρήσουμε τη γραμμή ότι υπάρχει ουδετερότητα και με τη νέα συμμετοχή και με τις νέες εξελίξεις. Δεν το λέω αυτό ότι αυτό θα ισχύσει για πάντα. Αυτό δεν μπορώ να το πω, αλλά στη φάση που βρισκόμαστε τώρα, ναι, ισχύει παντού. Σας ευχαριστώ κύριε Σκάλφιν. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Κυρία Υποψήφια Επίτροπε, η ασφάλεια για τον κυβερνοχώρο αποκτά μεγάλη σημασία. Η ανάπτυξη τεχνολογιών μέσω του διαδικτύου δημιουργούν αυξανόμενο κίνδυνο για τα κρίσιμα ε, δίκτυα για την ενημέρωση και πληροφόρηση των ε, πολιτών εν γέννη. Χρειάζεται διαφανείς ρυθμίσεις σε ασφάλεια του διαδικτύου και αποτελεσματική επιβολή. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να τύχει ισορροπία μέτρων για τη δημιουργία ασφαλούς κυβερνοχώρου και σεβασμού των θεμελιωδών δικαιωμάτων καταναλωτών ταυτόχρονα για να μην υπάρχουν καταχρήσεις. Θα είναι η ασφάλεια του κυβερνοχώρου στο πρόγραμμα στο μελλοντικό, κύριε Υποψήφιο Επίτροπε. Θα υπάρχει συντονιστής για την ασφάλεια του κυβερνοχώρου, μια θέση που υπάρχει στι ΣΥΠΑ και άλλε χώρες θα υπάρξει για την Ευρώπη. Τέτοιο συντονιστή μπορεί να συντονιστεί ίσω 27 εθνικού συντονιστέ ασφαλεία κυβερνοχώρου. Θα μπορέσετε να κάνετε τα δέατα ώστε να πετύχει διεθνή ε, συνεργασία με το... στον τομέα αυτό προχωρά πολύ γρήγορα η Ευρώπη. Απάντηση. Μας ενδιαφέρει πολύ αυτό που αναφέρατε. Είναι ένα από τα θέματα που δεν αφορά μόνο την κατάχρηση μιας καταστάσεως υπάρχει και ποινική πτυχή, εγκληματική πτυχή. Είναι κάτι παραπάνω επίθεση κατά των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αναφέρθηκα στο θέμα του Google. Αυτό που διάβασα το πρωί σε μία εφημερίδα αφορούσαν το έγκλημα στον κυβερνοχώρο που είχε σαν στόχο μία από τις μεγάλες τράπεζες. Οι πελάτες της τράπεζας έπαιρναν ηλεκτρονικό μήνυμα, email. Όπως μου είπα και από τα μέλη του γραφείου μου, και είναι σύμπτωση αυτή, μέλη του γραφείου μου πήραν email με ίδιο περιεχόμενο. Τι έλεγε, ότι η τράπεζά τους, έλεγε το email, φαινόταν ότι είναι γράμμα από την τράπεζά τους. Και έλεγε η τράπεζα υποτίθεται πρέπει να αλλάξει το σύνθημά σου, το password. Και πήγαινε σε ψευτό ιστοσελίδα που ήταν ακριβώς ίδια με την αληθινή Δίνεις εσύ τις λεπτομέρειες και από τη στιγμή που οι εγκληματίες δίνουν το password και λοιπά, το παίρνουν. Νομίζω ότι είναι η τραπεζά σου, το δίνεις στους εγκληματίες. Και είναι πολύ πιστική παγίδα και υπήρξαν πολλά θύματα. Ανησυχώ για τέτοιου είδους ε, επιθέσεις. Μου είπαν ότι υπάρχει και μαύρη αγορά, όπου οι εγκληματίες και οι hackers μπορούν να βρουν ιούς, διευθύνσεις email κλπ. Λεπτομέρειες σωστικών καρτών, ε, κωδικούς πρόσβασης κλπ. Πάνω από ένα εκατομμύρια ΙΗ εντοπίστηκαν το 2008 και το κόστος του εγκλήματος του κυβερνοχώρο αυξάνεται πολύ. Δεν περιορίζεται από σύνορα, είναι παγκόσμιο θέμα, οπότε αυτό που είπατε ότι χρειάζεται συνεργασία είναι πολύ λογικό. Διαφορετικά, απλώς ε, βλέπουμε πολύ μικρή περιοχή. Μία από τις προτεραιότητες μου για το πρόγραμμα το ψηφιακό θα είναι η Ευρώπη να είναι η ασφαλέστερη περιοχή στον κόσμο για τους καταναλωτές όσον αφορά το διαδίκτυο. Και ελπίζω όταν ρωτήσετε το δεύτερο ερώτημα να έχω τη δυνατότητα να επεκταθώ. Συμπληρωματικό ερώτημα. Ευχαριστώ. Επανέρχομαι στο θέμα αυτό για τον ε, τσάρο του κυβερνόχωρου ή τον συντονιστή του κυβερνόχωρου όπως τον λένε σε κάθε χώρα είναι άτομα τα οποία έχουν πραγματικά εξουσία να παρακολουθούν τι γίνεται στον κυβερνόχωρο και τι μέτρα θα πρέπει να ληφθούν για να αυξηθεί η ασφάλεια και είναι απαραίτητη η συνεργασία του σε διεθνέ επίπεδο. Θα θέσω και πάλι το ερώτημα. Θα είσαστε έτοιμοι να υποστηρίξετε να υπάρχει και ένα αρμόδιο για την κυβερνοασφάλεια μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και επίσης ε, τι συμβαίνει σε σχέση με την οδηγία για την ε, φύλαξη των δεδομένων, η οποία την χάνει κατάχρηση πάρα πολλέ φορέ. Στη Βουλγαρία η αστυνομία έχει σχεδόν απρόσκοπτη πρόσβαση σε πληροφορίε σε σχέση με την κινητή τηλεφωνία. Τι θα κάνετε λοιπόν για να έχετε αυτή την ισορροπία, από τη μια μεριά να υπάρχει η ασφάλεια στο, στο κυβερνόχώρο και να μην υπάρχει υπερβολική πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα. Λοιπόν, αυτό το οποίο αναφέρεται για <clears throat> την ε, οδηγία προστασίας των ε, δεδομένων είναι αρμόδια η κυρία Ρέντινγκ. Αυτή λοιπόν θα πρέπει να λάβει υπόψη αυτές τις πτυχές και να προχωρήσει σε ενδεχόμενη μεταρρύθμιση της οδηγίας. Πιστεύω και εγώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχουμε σαφείς θέσεις και να μην χρονοτριβούμε και να εργαστούμε όλοι για να αντιμετωπίσουμε τα θέματα αυτά και <clears throat> θα πρέπει και οι εμπλεκόμενοι στο δημόσιο και στο ιδιωτικό τομέα να συμμετάσχουν σε αυτό τον προβληματισμό. Αν με εγκρίνετε λοιπόν, αυτό το οποίο θα προτείνω θα είναι μια μείζον στρατηγική ενίσχυση τη ικανότητα τη Ευρωπαϊκή Ένωση σε ό,τι αφορά την ασφάλεια των πληροφοριών με ένα νέο ρόλο για το ΕΝΙΣΑ, το Ίδρυμα για την Ασφάλεια των Δικτύων. Κύριε Φύση, έχετε το λόγο. Γεια σας και καλημέρα και ευχαριστώ για την παρουσία σας κυρία Υποψήφια Επίτροπε δυστυχώς <coughs> οι πάροχοι υπηρεσιών δεν είναι πάντα ικανοποιημένοι με αυτά τα οποία προέκυψαν από την απελευθέρωση στην, ε, στις υπηρεσίες διαδικτύου. Τώρα έχουν στραφεί στη βραχυπρόθεσμη κερδοφορία λόγω της οικονομικής κρίσης. Επομένως, ορισμένες γεωγραφικές περιοχές δεν είναι αρκετά ε, ελκυστικές λόγω της γεωγραφικής τους ιδιαιτερότητας μέσα στο πλαίσιο αυτό. Και λαμβάνοντας υπόψη τις ε, κατευθυντήρες γραμμές για τις ε, κρατικές ενισχύσεις ενταχεία ανάπτυξη ευρυζωνικών υπηρεσιών που οδήγησαν στην ε, χρήση τέτοιων δικτύων. Αυτό πιστεύω ότι είναι ένα σημαντικό στοιχείο για να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα. Εσείς τι μέτρα προτείνετε να λάβετε για να δώσετε την ε, κίνητρα για την εφαρμογή δικτύων νέας γενιάς και να επιταχύνετε τη λειτουργία προγραμμάτων τα οποία ήδη είναι κινήσει και περιμένουν την έγκρισή σας. Έχω δύο γραμμές που μπορούμε να πάρουμε. Καταρχήν αυτές οι <clears throat> περιοχές της υπέθρου, αυτές οι περιοχές όπου δεν είναι ιδιαίτερα ελκυστικές για ιδιωτικούς επενδυτές, εκεί επιτρέπεται να υπάρχουν κρατικές επιδοτήσεις οι οποίες θα καλύψουν το κόστος με πρωτοβουλία του κράτους μέλους. Και επιπλέον υπάρχει η πρωτοβουλία της Κομισιόνου, η οποία αναλήφθη πέρσι η πρόπεση. Υπάρχουν τα απαραίτητα κονδύλια, αλλά δεν τα εκμεταλλεύτηκαν μέχρι στιγμής όλα τα κράτη-μέλη. και δεν επομένως προχώρησαν αρκετά τέτοια προγράμματα στον τομέα των ευρυζωνικών ψηφιακών υπηρεσιών για το άλλο τμήμα που αναφέρατε, όταν υπάρχει ενδιαφέρον των ιδιωτικών επενδυτών, θα πρέπει να συζητήσουμε, να κάτσουμε μαζί τους και να συζητήσουμε και σας ε, υπενθύμησα προηγουμένως ποια ήταν η δική μου εμπειρία ότι το να βρίσκονται σε μια στρογγυλή τράπεζα όλοι οι εμπλεκόμενοι στα θέματα αυτά μπορεί να οδηγήσει σε μια κατάσταση αμοιβαίω επωφελή για όλους. Και δεν πρέπει να είναι μονάχα οι ήδη εγκατεστημένοι στην αγορά, αλλά και οι νέοι νεοεισερχόμενοι στην αγορά που θα πρέπει να έχουν ίσες συνθήκες ανταγωνισμού και να έχουν και τη διαφάνεια και την νομική αρρωγή που είναι απαραίτητη. γιατί πολλές φορές θέλουν και αυτοί να ξέρουν ποιε είναι οι απόψει μας για το μέλλον και πώς υποστηρίζουμε το νομικό πλαίσιο το οποίο είναι απαραίτητο. Να ξέρουμε, είναι απαραίτητο για αυτού λοιπόν να υπάρχει ασφάλεια δικαίου, να ξέρουν ποια είδη ρυθμίσεων θα ισχύσουν για αυτούς. Είναι απαραίτητο λοιπόν να του τα εξηγήσουμε όλα αυτά. Ε, συμπληρωματικό ερώτημα, ναι κ. Ντέβιτ Σαν που ήταν προηγουμένω εκπρόσωπος του Γραφείου Ευρεσιτεχνιών στην, ε, στο φορέα της Ευρωπαϊκής Ένωσης έλεγε ότι αν δεν υπήρχε ένα σύστημα αν υπήρχε ένα σύστημα ενιαίο σε ευρωπαϊκό επίπεδο θα μπορούσε με τον τρόπο αυτό να αρθεί η πολυμορφία των ε, ευρωπαϊκών συστημάτων έγκριση Ευρεσιτεχνιών. Για τα φαρμακευτικά προϊόντα δημιουργήθηκε κατά κάποιο τρόπο ένα τέτοιο ενιαίο σύστημα για να υπάρξει μια νομολογία ευρωπαϊκού χαρακτήρα. Συμφωνείτε λοιπόν με την άποψη του κυρίου Ντέβιτ Σάντ και αυτή είναι μια άποψη που ακολουθούν και οι μεγάλε πολυεθνικέ εταιρείε λογισμικού. Είναι απαραίτητο να υπάρξει ένα ευρωπαϊκό <clears throat> δικαστήριο κατά κάποιο τρόπο για τι ε, ευρεσιτεχνίε. Είναι συναρπαστικό ερώτημα. Καταρχήν όμως δεν είναι θέμα του χαρτοφυλακίου μου, αλλά το γραφείο έβρεση τεχνιών κάνει θαυμάσια εργασία και αυτό το έργο θα πρέπει να γίνει σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Πάντως θα πρέπει να διασαφινιστεί αν αυτό είναι ο καλύτερος δρόμος για τις ευρεσιτεχνίες και το λογισμικό, γιατί το μεγαλύτερο πρόβλημα με τη Microsoft ήταν η διαλειτουργικότητα και την προηγούμενη εβδομάδα <clears throat> καταφέραμε να έχουμε μια τελική συμφωνία. Η διαλειτουργικότητα για τα λογισμικά είναι πολύ καλύτερη πλέον προς το συμφέρον της οικονομίας και του καταναλωτή. Τώρα, αν υπάρχουν ακόμα θέματα αβεβαιότητος όπως τα είδη των προτύπων τα οποία θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν, εκεί θέλω να είμαι λιγάκι επιφυλακτική. Αλλά το σημείο αυτό θα επανέλθει και θα πρέπει να συζητήσουμε τι θα πρέπει να γίνει με τις ευρεσιτεχνίες στον τομέα του λογισμικού και θα ήθελα να έχω και τις δικές σας απόψεις για το θέμα αυτό. οι συνάδελφοι από την Επιτροπή Πολιτισμού, η πρόεδρος της Επιτροπής Πολιτισμού, η Δόρη Πακ. Κυρία Κρούς, εδώ και χρόνια αγωνιζόμαστε στην Επιτροπή Πολιτισμού για να υπάρξει ένα ευρωπαϊκό μοντέλο ρύθμισης για τις ραδιοσυχνότητες. Γιατί αυτό είναι η καλύτερη εγγύηση για την εκπαίδευση και την έκφραση, την ελεύθερη των, των απόψεων. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να υπάρχει ένα σύστημα το οποίο είναι ουδέτερο προ την τεχνολογία και επιτρέπει ένα ανοιχτό δημόσιο ραδιόφωνο. Κατά την άποψή σα, ποιο είναι ο ρόλο που πρέπει να παίξουν οι δημόσιε υπηρεσίε στον τομέα των μέσων ενημέρωση. Κύριε Κρούζ, μια σαφή ερώτηση. Είναι σαφής ερώτηση. Ξέρουμε ότι ανάλογα με τις δημόσιες υπηρεσίες εκπομπών αναμετάδοσης προσπαθούμε να τηρούμε τις ίδιες αρχές παντού και προσπαθούμε να έχουμε και ξεχωριστές ε, λύσεις προσαρμοσμένες αλλά θα πρέπει να είμαστε σαφές ότι ο ορισμός θα πρέπει να είναι ξεκάθαρος. Ιδάλλως δεν θα προκύψει πραγματικό αποτέλεσμα από τις συζητήσεις μας. Και αυτό που κάναμε στο παρελθόν στον ανταγωνισμό, σε θέματα ανταγωνισμού. Φαντάζομαι ότι σας ε, βρήκε και σας σύμφωνους για να ανταποκριθούμε στην πολυμορφία που εξακολουθεί να υφίσταται και αποτελεί το μεγάλο θέμα. Ένα από τα θέματα που μας απασχολεί στην Ευρώπη, αλλά παράλληλα να υπάρχει και μια ανταγωνιστική αγορά στην οποία στην τελική ανάλυση ο καταναλωτής θα μπορέσει να διαλέξει αυτό που προτιμά. Δεν ικανοποιήθηκε στην απάντηση, αλλά να ρωτήσω και, να ρωτήσω και κάτι άλλο για την, ε, την ε, UNESCO. Ήσασταν κατά της, ε, τον δεσμευτικού χαρακτήρα της συνθήκης αυτής της UNESCO. Έχετε αλλάξει πλέον γνώμη. Πιστεύετε ότι με το μέσο αυτό μπορούμε να προωθήσουμε την ε, παράδοση του πολιτισμού και της πληροφορίας στην Ευρώπη. Απάντηση. Δεν, ε, ξέρω τι υπήρχε, δεν ήξερα ότι υπήρχε τέτοια διαφοροποίηση, αλλά αν με ρωτάτε κατά πόσο στο συγκεκριμένο χαρτοφυλάκιο και σε ό,τι αφορά τον πολιτισμό και τη σχέση του με το θέμα που διαπραγματευόμαστε εδώ, θεωρώ ότι είναι απόλυτα απαραίτητο να υπάρχει σαφήνεια. Ιδιαίτερα χάνουμε, γιατί αλλιώς χάνουμε ευκαιρίες και υπάρχουν πραγματικά τεράστιες ευκαιρίες στην ψηφιακή ατζέντα, τις οποίες θα πρέπει να αξιοποιήσουμε. Κυρία Κάμεραβερτ, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κυρία Κρούς, έχουμε ένα πακέτο για τις τηλεπικοινωνίες όπου αναφέρουν μια σειρά από αρχές που λέει ότι το, ψηφιακό, το λεγόμενο ψηφιακό μέρισμα πρέπει να γίνεται προς το καλό και της οικονομίας αλλά και, των, και της κοινωνίας και επίσης ότι πιστεύουμε στον πληροφορισμό των μέσων ενημέρωσης και στην πληροφορία, την πολυμορφία της ε, πληροφόρησης. Αλλά το έγγραφο το οποίο έχουμε τώρα από την Κομισιόν, αυτές τις αρχές που έχουν να κάνουν με την πολιτική ραδιοσυχνοτήτων δεν αναφέρονται καθόλου. Μονάχα οι οικονομικές πτυχές είναι αυτές οι οποίες έχουν την πρωτοκαθεδρία. Γι' αυτό θέτω το εξή ερώτημα. Συμφωνείτε ότι για την κινητοποίηση του ψηφιακού μερίσματος θα πρέπει να ληφθούν όχι μόνο οικονομικές προδιαγραφέ, αλλά και κοινωνικές και πολιτιστικέ, και αν ναι, πώς θα ξέρετε την κατάλληλη ισορροπία μεταξύ αυτών των αντιμαχωμένων ε, συμφερόντων στον τομέα αρμοδιότητό σα. Ενδιαφέρον θέμα τίθεται εδώ, όπου και εδώ συμμετέχουν κατά πολύ τα κράτη-μέλη και συζητείτε τι αντιμετωπίζουμε με τις νέες συνέπειες του κανονιστικού πλαισίου που δεχθήκατε. Θα πρέπει να ληφθεί υπόψη και θα είναι αποτυχία αν απλώς βγάλουμε εκτός τον πολιτισμό ή τα μέσα ενημέρωσης. Πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι είναι ένας από τους ε, εμπλεκομένους Υπάρχει δυνατότης, αλλά δεν θα πρέπει να ακολουθηθεί εντελώς διαφορετική μεταχείριση. Ευχαριστώ. κυρία Κρούς. Θα ήθελα να υπάρχει όμως μια ισορροπία μεταξύ των οικονομικών ε, συμφερόντων και των πολιτισμικών και πολιτιστικών στοιχείων. Αλλά έχω να κάνω και μια άλλη ερώτηση για τη συχνότητα γιατί όταν οι εδαφικές συχνότητες είναι σαφές ότι θα αποτελέσουν ε, σημαντική τεχνολογία και για την ε, ραδιοεκπομπές. Πώς θα διασφαλίσετε λοιπόν ότι και αυτή η εδαφική πλατφόρμα θα συνεχίσει να διατίθεται και θα διασφαλιστεί το γενικό συμφέρον χωρίς να προαχθεί ειδικά το οικονομικό συμφέρον εις βάρος των άλλων ε, στοιχείων απάντηση. Άκουσα τι είπατε και αναφέρθηκα προηγουμένως, δεν θυμάμαι σε ποιον βουλευτή, σε έναν από τους συναδέλφου σας, ότι θα πρέπει να υπάρχει ουδετερότητα του δικτύου, θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα κατά την οποία οι εδαφικές, ε, δορυφορικές και καλωδιακές συνδέσεις θα την χάνουν με ταχύρισης, με τρόπο ο οποίος θα τους επιτρέψει να αναπτυχθούν ως προς τις υπηρεσίες τους. Άρα μην ανησυχείτε, δεν πρόκειται να παραμεριστούν αυτές οι υπηρεσίες. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος, ο κ. Καβαντά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κυρία μου, δεχόμαστε θετικά την ε, δήλωσή σας. Έχετε ένα ερωτηματικό ε, στην μπουτονιέρα σας, στην καρφίτσα Εγώ έχω στο κεφάλι μου ένα ερωτηματικό. Εδώ Μιλάμε βιομηχανία, επενδύσεις, συστήματα, σωλήνες κλπ. Ρυθμίνης. Δεν μιλάμε για περιεχόμενο. Οδηγούμε θα δικαιωθούμε προς μεγάλη καταστροφή αν αφιερωθεί η θητεία σας μόνο στην διοργάνωση των ψηφιακών βιομηχανιών, διότι χωρίς περιεχόμενο δεν θα πετύχουμε πολλά και τα περιεχόμενα προέρχονται από αλλού. Δηλαδή, είμαστε στην περίπτωση εκείνων που είναι αντικείμενο εκμετάλλευση περισσότερο, παρά εκμεταλλεύω το θέμα. Όπω είπε και ο πρόεδρο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ε, έχετε ευθύνη για τρία-τέσσερα θέματα που ενδιαφέρουν πολύ. Πώ θα εργαστείτε αποτελεσματικά, πρώτα απ' όλα με τις την πολιτιστική βιομηχανία, τα πνευματικά δικαιώματα και του κανόνε που ε, εφαρμόζονται όσον αφορά την κατανάλωση αγαθών και πολιτιστικών αγαθών Πώς θα λειτουργήσει στα πλαίσια του συντονισμού με τους άλλους επιτρόπους που πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής διασκόρπισε και αυτό είναι λάθος και δημιουργεί ε, δυσκολίες αυτό. Η κυρία Κρούσια να απαντήσει. Δεν θα με κατηγορήσετε εάν δεν εκφράσω τις σκέψεις μου για το τι θα ήταν καλύτερο για να, το έχει, να έχει κανείς ένα χαρτοφυλάκιο. Ο πρόεδρος έκανε πολύ καλή δουλειά, ήταν επιτυχής διότι έδωσε 26 υποψήφιου ε, επιτρόπους ένα χαρτοφυλάκιο το οποίο να αξίζει τον κόπο. Αυτό δεν μπορούσε να. δεν ήταν εύκολο και δεν είναι μυστικό αυτό που λέω. Τώρα και 26 έχουν ένα χαρτοφυλάκιο και κατά κάποιο τρόπο κάποια χαρτοφυλάκια χάνανε κάποιο μερίδιο συγκρίση με άλλα. Εν γέννη η δουλειά ήταν έξοχη αυτή που έγινε. Είναι ένα σύστημα συνεργασίας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παίρνει στο τέλος την απόφαση. Ποτέ ένας επίτροπος μπορεί να πει εγώ πήρα αυτή την απόφαση γίνεται δεκτή μια πρόταση μόνο όταν υποστηρίζεται από όλη την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, από το σώμα. Αυτό είναι το όφελο της πενταετού εμπειρία. Αυτό το συλλογικό πνεύμα στις περισσότερε περιπτώσεις είναι κάτι πολύ θετικό. Ήθελα να το πω και στην εισαγωγική μου ομιλία αυτό. Όσον αφορά αυτό το χαρτοφυλάκιο, Πρέπει να υπάρχει πολύ καλή επαφή με τον Μισελ Μπαρνιέ, με την κυρία Αντρούλα Βασιλείου, ξέρω μόνο τα μικρά ονόματα. Τέλο πάντων με τον Γιάννη Πατότσνικ, με τη Βιβιά, Μόρα Γκέγκεν Χουίν επίσης. Είναι πρόκληση αυτή ότι πρέπει να συζητούμε περισσότεροι από δύο καμιά φορά, καμιά φορά μόνο δύο, να συζητούμε συγκεκριμένα θέματα. Συνεργασία είναι το σημαντικό. Αν δεν επικρατεί η σωστή το σωστό συλλογικό πνεύμα, έχετε δίκιο, αλλά ο Μπαρόσο θα επιτηρεί. Και αν υπάρχει κάποια τριβή ή κάποιος καυγάς, κάποια προβλήματα θα παρέμβει. Εγώ είμαι, ο χαρακτήρας μου είναι να θέλω να εργάζομαι ομαδικά και μου αρέσει πολύ να ανήκω σε ομάδα. Ο κύριος Καβαδά για την ε, δεύτερη ερώτηση. Έχω συμπληρωματική ερώτηση που βασίζεται λίγο σε αυτά που είπε η κυρία Ντόρις Πακ. Θα μπορείτε να μας πείτε, κυρία μου, εδώ και 20 χρόνια αναπτύξαμε τα ιδιωτικά μέσα στην Ευρώπη με μεγάλη επιτυχία, όμως έχει ε, επιδεινωθεί πολύ η ποιότητα και η ενημέρωση των πολιτών. Θα είσαστε υπέρ βοηθείας των δημοσίων ραδιοφώνων και τηλεοράσεων όταν υπάρχουν βρίσκονται σε θέση ελλείψης οροπίας σε δυσχερή θέση έναντι των ιδιωτικών ε, καναλιών και ραδιοφωνικών σταθμών. Δηλαδή τελικά να υπάρχει μια ισορροπία και γίνεται σεβαστή. Μ' αρέσει η ποικιλομορφία λέει ο κυρία Κρούς. Βεβαίως ενδιαφέρομαι πολύ για την ποιότητα και από την πλευρά του δημόσιου, των δημοσίων μέσων και των ιδιωτικών τα δημόσια μέσα έχουν ακόμα μεγαλύτερη ευθύνη όσον αφορά την ποιότητα που πρέπει να συμπεριλαμβάνουν. Διότι έχουν ειδικό καθήκον και στόχο. Αλλά προσπαθήσουμε να καλύψουμε και τα δύο. Θέλουμε ισορροπία, ναι. Η γλώσσα του σώματός σας είναι η γλώσσα του δικού μου σώματος. Και ας μην μιλάμε. Πιστεύω ότι πρέπει να έχει ισορροπημένο σύστημα. Ίσες ευκαιρίες και το προϊόν είναι τελικά αυτό που αντιστοιχεί στον πολιτισμό μας, στην κουλτούρα μας, στους πολίτες μας και στην οικονομία μας. Γιατί και αυτό είναι ένα κομμάτι της οικονομίας. Κυρία Τούν Χόενστάιν, κυρία Επίτροπε, για να συνεχίσω τα ερωτήματα που έθεσε, έθεσαν οι συνάδελφοί μου από την Επιτροπή Πολιτισμού. Μιλήσαμε για το ράδιο, ραδιόφωνο ποια είναι τα προβλήματα που έχουν να αντιμετωπίσουν οι, οι συντάκτες εντύπων στο ίντερ, ε, από το ίντερνετ. Έχουν πρόβλημα ανταγωνισμού. Αλλάζουν ε, την ε, κερδοφορία των εντύπων τους. Μειώνουν την ποιότητα και υπάρχουν πολλοί οι οποίοι βρίσκονται σε μειονεκτική θέση, ενώ άλλοι εκμεταλλεύονται το, το περιεχόμενο που βρίσκεται και στο διαδίκτυο μαζί με το έντυπο περιεχόμενο για εμπορικούς στόχους, κάτι το οποίο μπορεί να γίνει σήμερα με την ταχεία ανάπτυξη της τεχνολογίας. Ποια είναι η πρότασή σας να για να δημιουργήσουμε ένα σύστημα το οποίο θα δώσει πρόσβαση σε ευρύ περιεχόμενο για τον πελάτη, για τον ε, καταναλωτή, αλλά δεν θα θέσει σε κίνδυνο το τα συμφέροντα των συντακτών εντύπων μέσων και, θα, και των καταναλωτών και θα ενθαρρύνει συγχρόνως την ανάπτυξη της ε, τεχνολογίας της πληροφορίας. Number one, two. Πρώτα απ' όλα, να δώσουμε έναυσμα για όλους να γνωρίζουν ότι αν παραμείνουν στην οδηγό γραμμή που έχουν μέχρι τώρα δεν θα υπάρξει καμία λύση. Θα πρέπει να συνδυάσουμε την παραδοσιακή τους παροχή πληροφοριών με τα νέα μέσα για να έχουμε τη δυνατότητα να παρέχουμε πληροφορίες και με τα νέα μέσα ενημέρωσης. Πιστεύω σε μια ανταγωνιστική αγορά όπου θα πρέπει να έχουν την ευκαιρία να το πράξουν αυτό. Συμπληρωματικό ερώτημα. Αν μιλάμε για τις ευκαιρίες οι οποίες παρέχονται από την αγορά και αν μιλάμε για την αρχή της μη διάκρισης θα είσαστε τόσο σκληροί όσο υπήρξετε με ορισμένε από τι αποφάσει σα ω ε, Επίτροπο Ανταγωνισμού. Εγώ είμαι από την Πολωνία, όπω ξέρετε. Θα είσαστε αρκετά σκληροί για να εξασφαλίσετε ότι εφαρμόζεται η αρχή της μη διάκριση για όλους τους Ευρωπαίους πολίτες οι οποίοι χρησιμοποιούν τη δυνατότητα αγορών στο διαδίκτυο. Δεν υπάρχει ίδια προ... πρόσβαση σε όλους. Ένα από τα παραδείγματα είναι η μουσική από το iTunes. Ποιε θα είναι οι επόμενε δράσεις σα για να εξασφαλίσετε ότι όλοι έχουν πρόσβαση σε τέτοιες υπηρεσίε. Δεν σκέφτηκα να αλλάξω το χαρακτήρα μου. Επομένως, ακριβώς αυτό το οποίο περιμένετε σε επίπεδο αυστηρότητος θα υπάρχει. Εγώ είμαι διάφανη, είμαι ε, προβλέψιμη και προσπαθώ να είμαι δίκαια. Επομένως αυτό μπορείτε να το λάβετε υπόψη σε όλες τις συζητήσεις οι οποίες θα ακολουθήσουν. Όταν ασχολείστε με τα θέματα των αγορών ε, <clears throat> στο διαδίκτυο. Αυτό το ζήτημα ήταν ένα από αυτά τα οποία ήταν για μένα κυριότερος λόγος να αντιμετωπίσω τα θέματα αυτά της μουσικής στο διαδίκτυο μέσα σε αυτό το στρογγυλό τραπέζι με όλους τους εμπλεκομένους. Το αποτέλεσμα ήταν ότι στην τελευταία μας συνάντηση με τους εμπλεκόμενους για τα θέματα αυτά, με τους κυρίους αυτούς και κάποιες κυρίες στην στρογγυλή αυτή τράπεζα, συμφωνήσαμε σε μια σειρά αρχών και εγώ είμαι υπερήφανη που κανείς δεν είχε αποχώρησε από αυτή την ομάδα και δεν είχε αντίρρηση. Τελικά καταλήξαμε σε μια συμφωνία. Τώρα όμως ερχόμαστε στη φάση της εφαρμογής και αυτή θα είναι δύσκολη. Να είσαστε σίγουροι όμως ότι εγώ θα κάνω ό,τι είναι ανθρωπίνως δυνατό για να επιτύχουμε την σωστή εφαρμογή. Εγώ δεν μπορώ πραγματικά να εξηγήσω γιατί στην Πολωνία ή σε κάποια άλλη χώρα δεν μπορεί κανείς να κατεβάσει από το διαδίκτυο, αυτό μπορεί να κατεβάσει σε άλλα κράτη που βρισκόνται σε μια ενιαία αγορά. Η κυρία Χάνιμπαλ. Ευχαριστώ πρόεδρε κυρία Κρούς. Θα ήθελα να επανέλθω στο θέμα που αναφέρατε και προηγουμένως για το περιεχόμενο και την ποιότητα. Ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τον πλουραλισμό των μέσων, το οποίο είναι ένα θέμα στο Κοινοβούλιο, το οποίο έχουμε διαπραγματευτεί και φαίνεται ότι αυτή η προσέγγιση τριών επιπέδων που έχουν το 2007 και μετά δεν ήταν πολύ αποτελεσματική και αυτό μάλιστα σε μεγαλύτερο βαθμό σε κάποια, σε κάποια κράτη-μέλη και κινδυνεύουμε να χάσουμε και άλλο ποσοστό της πολυμορφίας των μέσων σε ό,τι αφορά θέμα πολιτικό, θέματα πολιτικά, πολιτισμικά και περιεχομένου. Θα ήθελα λοιπόν να μας πείτε τι συγκεκριμένες δράσεις θα πάρετε για να διασφαλίσετε ότι θα προωθηθεί ο πλουραλισμός των μέσων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Απάντηση. Το να φέρουμε σε επαφή τα εμπλεκόμενα μέρη, να εντοπίσουμε πού είναι το πρόβλημα, ποια θα μπορούσε να είναι μια ενδεχόμενη λύση και στη συνέχεια να προσπαθήσουμε να βρούμε έναν τρόπο να βρούμε τις λύσεις αυτές και να τις ακολουθήσουμε. Είναι πολύ σημαντικά όλα αυτά για τον πλουραλισμό των μέσων όχι μόνο για σας αλλά και για μένα. Για να επανέλθω, θεωρώ ότι είναι δύσκολη η πρόκληση αυτή, γιατί κάποια από τα άτομα που συμμετέχουν είναι γνωστό ότι δεν θέλουν να μιλήσουν με κανέναν. Ίσως λοιπόν θα χρειαστεί να ακολουθήσουμε πιο σκληρή στάση, αν θέλουμε στα σοβαρά να προωθήσουμε αυτή την πολυμορφία. Σε ό,τι αφορά τα εθνικά και ευρωπαϊκά μέσα και τις ειδήσει. Απάντηση, δώστε μου μια ευκαιρία. Ξέρω φυσικά ότι είναι δύσκολη αυτή η πρόκληση, δεν υπάρχει αμφιβολία. Αλλά θεωρώ ότι έχω αντιμετωπίσει και στο παρελθόν δύσκολε καταστάσει. Αφήστε με να φέρω σε επαφή τα διάφορα μέρη για να εντοπίσουμε ποιο είναι το πραγματικό πρόβλημα. Κατά πόσο βγάζει νόημα, κατά πόσο υπάρχει μία λύση, κατά πόσο μπορεί να εξευρεθεί κάποιος συμβιβασμός. Αλλά σε κάθε περίπτωση θα επιδιώξουμε ένα σαφές αποτέλεσμα. Αν δεν το καταφέρουμε αυτό, ασφαλώς και θα αναλάβουμε δράση. Αυτό δεν τίθεται σε συζήτηση. Ο Πρόεδρος, ευχαριστώ. Κυρία Σχάκε. Ευχαριστώ, Πρόεδρα, και καλωσορίζω την Επίτροπο. Μας δώσατε με σαφήνεια το όραμά σας και ακούσαμε και πολλές ερωτήσεις και απαντήσεις. Μιλήσατε για την τεχνολογία, την ανάγκη διαφόρων υποδομών, αλλά μιλήσατε και για τον αντίκτυπο στην δημοκρατία και στην κοινωνία αναφορικά με την ψηφιακή ατζέντα ήρθα σε επαφή με κάποιους πολίτες και θα σας θέσω λοιπόν μια ερώτηση την οποία που μου έθεσαν μέσω υπολογιστή κατά τη διάρκεια πριν από την ακρόαση αυτή για να δείξω ότι υπάρχει και εισερχόμενη ροή. Να σας θέσω το ερώτημα του Μάρκ λοιπόν, ο οποίος λέει ότι συνεργάζεστε με πολλούς συναδέλφους στο χαρτοφυλάκιό σας, το οποίο εμπλέκει διάφορους τομείς. Θα συνεργαστείτε και με τη Λέδη Άστον τον υποψήφιο Επίτροπο Φιούλε και άλλους ε, επιτρόπους υποψήφιους για να διασφαλίσετε ότι θα εξασφαλιστεί η ελευθερία της έκφρασης σε ό,τι αφορά την ψηφιακή ατζέντα και ότι θα τεχθεί στην πολιτική της Ένωσης. Είμαι πάρα πολύ ευγνώμων για αυτή την ερώτηση του Μάρτ. Δεν είναι εύκολη η ερώτηση βέβαια. Η απάντηση μπορώ να δώσω από το βάθος της καρδίας μου και θα κάνω ό,τι μπορώ περισσότερο είναι γεγονός ότι η κάθε Άστον ενδιαφέρεται ιδιαίτερα για την ελευθερία της ε, έκφρασης και για πολλά άλλα θέματα. Σίγουρα θα θίξω αυτό το ζήτημα και με τον κύριο Φίλε. Αυτό είναι το πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι αυτού του χαρτοφυλακίου, διότι συνδέει διάφορους τομείς του επιστητού. θα ήταν πιο εύκολο να σας πω ποιοι δεν εμπλέκονται στα θέματα τα ψηφιακά. Και δεν μπορώ να σκεφτώ να υπάρχει και κάποιο αρτοφυλάκιο που δεν έχει κάποια σχέση με αυτά. Ευχαριστώ. Εδώ εκπροσωπώ την Επιτροπή Πολιτισμού Μέσων Ενημέρωσης και Παιδείας και φυσικά η ελεύθερη καλλιτεχνική δημιουργία είναι πάρα πολύ σημαντική για την Επιτροπή μας και μια σημαντική πηγή περιεχομένου που τώρα μπορούμε να διαδίδουμε στο διαδίκτυο και να δημιουργούμε και στο διαδίκτυο. Θα ήθελα να ξέρω από εσά λοιπόν Πώς βλέπετε αυτήν την συνεργασία μετά από την ε, ε, πολύ πιθανή έγκρισή σας από την Επιτροπή μας και πώς βλέπετε το θέμα αυτό της ε, ελευθερίας των μέσων κτλ. Είναι κεφαλαιόδες στον τομέα αυτό να εκμεταλλευτούμε όλες τις δυνατότητες οι οποίες ανοίγονται μπροστά μας και να αντιμετωπίσουμε όλες τις προκλήσεις. Και γι' αυτό, αυτό και για πολλούς λόγους. Στις περιπτώσεις αυτές που αναφέρω σας στο εκπαιδευτικό τμήμα των μέσων ενημέρωσης, οι νέοι, ακόμα και αυτοί οι οποίοι βρίσκονται στην διαβίου μάθησης, οι περισσότεροι είναι νέοι στη σκέψη τους, ούτως είπε. Εάν ισχύει αυτό λοιπόν, θα ήταν γελίο να μην χρησιμοποιήσουμε όλες τις ευκαιρίες για να προωθήσουμε αυτή την εκπαίδευση. Η γέφυρα λοιπόν αυτή προς την κουλτούρα υπάρχει και είναι σημαντικό επίσης μέσω της κουλτούρας να εξασφαλίσουμε μεγαλύτερη συμμετοχή από αυτούς που ενδιαφέρονται για τα πολιτιστικά θέματα, να καταλήξουμε σε μια αμοιβαίω υποφελή κατάσταση για να θίξουμε τα ζητήματα τα οποία αναφέρατε. Είναι θέμα καινοτροπίας. όταν μιλάμε για το έγκλημα Είναι θέματα τα οποία ενδιαφέρουν τους νέους, αλλά ακόμα και τους παλίμπεδες. Πολλές φορές δεν ξέρουν τι ακριβώς συμβαίνει με τα ιδιωτικά της στοιχεία και τις πληροφορίες που παίρνουν. Πρέπει λοιπόν να το θίξουμε αυτό το θέμα όταν μιλάμε για παιδεία και κουλτούρα. Και επομένως Μπορούμε να πούμε στους νέους, προτού βγάλετε κάτι στο διαδίκτυο, προσπαθήστε να επικοινωνείτε κιόλας. Εγώ δεν θα ανησυχούσα λοιπόν πάρα πολύ, γιατί πολλές φορές παίρνουμε πληροφορίες οι οποίες είναι άχρηστες. Ο Μάλκολμ Χάρμπορ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ήθελα να πάω στο βασικό σας χαρτοφυλάκιο κύριε υποψήφια επίτροπε. Εδώ είμαι, εδώ είμαι. Δηλαδή, πολλοί ανταγωνιστική αγορά τηλεπικοινωνιών που θα ενθαρρύνει τι επενδύσει. Και όπως είπαν αρκετοί συνάδελφοι, είσαστε πασίγνωστοι ω πρωταθλήτη, αν θέλετε, του ανταγωνισμού, προασπίζετε τον ανταγωνισμό και όποτε υπήρχαν θέσει στην αγορά τις αντιμετωπίζατε σε πολλού τομεί. Όπω τα γνωρίζετε, είμαι σίγουρο, το μέσο μερίδιο τη αγορά των ιστορικών εταιριών τηλεπικοινωνιών στην Ευρυζωνική στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι 45%. Και αυτό έτσι ήταν επί τρία χρόνια, τελευταία τρία χρόνια. Σε μια σημαντική αγορά έχουν ένα μερίδιο 57%. υποψήφια επίτροπε συμμερίζεται τη δική μου άποψη. Δηλαδή, αυτά τα υψηλά μερίδια της αγορά θα εμποδίσουν ανταγωνισμό και επενδύσεις. Και τι προτείνετε να κάνετε περί αυτού. Απάντηση. Είναι ένας λόγος να παρακολουθούμε αυτές τις καταστάσεις πολύ προσεκτικά και με αυστηρότητα μεγάλη. Διότι δεσπόζουσα θέση δεν σημαίνει ότι είναι κάτι απαράδεκτο. Εξαρτάται από τον τρόπο της συμπεριφοράς. Αν η δεσπόζουσα επιχείρηση συμπεριφέρεται με συγκεκριμένο τρόπο. Και όπως πανέφερα είχαμε παραδείγματα ε, διαφόρων κατηγοριών που συνέβαιναν αυτά. Ξέρω ότι κάποιες από τις παραδοσιακές επιχειρήσεις έχουν υψηλό μερίδιο της ε, αγοράς. Όμως, αν αυτό δεν πάει καλά, πρέπει να δράσουμε και χρειαζόμαστε στοιχεία. Και ο καθένας μπορεί να χτυπήσει την πόρτα μου για να αναφέρει. Ήλπιζα ότι θα ήσασταν ε, πιο τολμηροί σε αυτό, λόγω του παρελθόντος σας. Νομίζω ότι ήταν πολύ αδύναμη απάντηση, αν επιτρέπετε να το πω αυτό. Ποια είναι η απόψή σα λοιπόν για λειτουργικό διαχωρισμό, κάτι που ισχύει στη χώρα μου και στη χώρα που ξέρετε καλύτερα εσεί, στην Ολλανδία, όπου η KPN που είναι παλιά εταιρεία εγκαθιστά ανοιχτά δίκτυα για να αυξήσει τη ζήτηση για υπηρεσίε υψηλή ταχύτητα. Αυτού του είδου τα φάρμακα θα έπρεπε να προωθείτε εσεί για να αντιμετωπιστούν ε, τα, οι επιχειρήσει που έχουν πολύ μεγάλο μερίδιο, διότι όλα αυτά τα στοιχεία και θα έρθουν και άλλα σύντομα, τα στοιχεία δείχνουν ότι αυτός ο τρόπος είναι να προωθήσουμε τις ε, επενδύσεις και τον ανταγωνισμό. Απάντηση. Φαίνεται να υπήρξε κάποια παρεξήγηση, κύριε Πρόεδρε. Λέει η κυρία Κρούς. Ήμουν δραστήρια σε αυτόν τον τομέα πολιτικής ανταγωνισμού, αναμφισβήτητα. Έκανα τη δουλειά μου ούτως υπήν. Τούτου λεχθέντος, εμείς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν επετέθημεν κατά μερών που ήταν δεσπόζοντα και συμπεριφερόταν με κάποιο τρόπο. Ήμασταν διαφανείς όταν κινούμεθα κατά και όταν ζητούσαμε διορθωτικά μέτρα ή όταν λέγαμε απλώς όχι. Όσον αφορά τη λειτουργικό διαχωρισμό, κάναμε το ίδιο, το, κάθαμε, το κάναμε στον τομέα της ενέργειας, άρα πρέπει να είστε σίγουρος ότι αν κάποια δεδομένη στιγμή σε αυτό το τομέα μου δώσετε την ευκαιρία να δράσω Εάν υπάρξει κατάχρηση θα ε, δράσω. Κυρία Κορχόλα, ευχαριστώ. Κυρία Υποψήφια Επίτροπε, καλωσορίζω τα θετικά σας σχόλια που αναφέρατε στην ανάγκη για μια νέα αγορά στο ψηφιακό τομέα. Να προχωρήσω πιο πέρα με ένα συγκεκριμένο ερώτημα. Θα υποστηρίζατε την ιδέα ανεξάρτητα της ε, συστήματος βαθμολόγησης που θα ανανεώνεται κάθε χρόνο όσον αφορά την αγορά αυτά και θα γίνεται αξιολόγηση των κρατών μελών και τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω σύμφωνα με συγκεκριμένα αριθμιστικά κριτήρια για την ενιαία αγορά τη ψηφιακή. Απάντηση. Είμαι υπέρ αυτή τη προσέγγιση. Δώστε μου λίγο χρόνο, όχι σήμερα, να το σκεφτώ διεξοδικά το θέμα. Έχω την εμπειρία αυτού του συστήματος βαθμολόγηση. scoreboard, για τις κρατικές ενισχύσεις. Τομέας που είναι στην ευθύνη μου τώρα. Και εκείνοι που δεν ήταν θετικοί στην αρχή τελικά επίστηκαν. Είναι θετικοί σήμερα σε αυτό το σύστημα. δεν πιστεύω να υπάρχουν τώρα συζητήσει αν λειτουργήσε αυτό σε έναν τομέα ότι εδώ θα λειτουργήσει. Ευχαριστώ για την ανοιχτή σα τάση λέει η κυρία Καοχόλα, τι άλλες εναλλακτικές λύσεις θα μπορούσε να προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το ώστε να ολοκληρωθεί η ενιαία ψηφιακή αγορά το ταχύτερο δυνατόν. Απάντηση. Να είστε βέβαιοι ότι έχουμε το 2020, πρόγραμμα για το 2020 αυτής της Επιτροπής. Ο πρόεδρος Μπαρόσο υποστηρίζει αυτό το αυτή την προσέγγιση. Και από τα αγαπημένα του θέματα είναι αυτό το ψηφιακό πρόγραμμα, ψηφιακή ατζέντα. Και είναι σαφέ τι θέλει. Είναι από τα αγαπημένα του παιδιά. Λοιπόν, α προχωρήσουμε. Σε συνεργασία μαζί σα με τα κράτη-μέλη, σε συνεργασία με όλου του εμπλεκόμενου, εθνικού, ρυθμιστικού φορεί, όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, αν συνεργαστούμε μπορούμε να προωθήσουμε πολύ το όλο ζήτημα. Σας ευχαριστώ. Η κυρία Κούτσε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κυρία Κρούς, είμαι στα αριστερά σας. Στην αρχική σας παρέμβαση αναφερθήκατε στις ε, τεχνολογίες πληροφορίες που πρέπει να είναι προς την υπηρεσία του πολέτη. Αυτά μας οδήγησαν στο διαδίκτυο που συνδέει πολίτες με πολίτες, πολίτες με επιχειρήσεις κτλ. Και έχουμε ήδη τον κίνδυνο αυτό να έχουμε στο μέλλον συνδέσεις όχι με ανθρώπους, μεταξύ ανθρώπων, αλλά μεταξύ ανθρώπων και αντικειμένων, avatars στο ίντερνετ. Και το πρόβλημα σε αυτές τις περιπτώσεις είναι ότι δεν μπορεί να υπάρξει πλήρης προστασία τη ιδιωτική ζωή των πολιτών. Πώς, τι θα κάνετε για να εξασφαλιστεί αυτή η προστασία. Αυτό είναι ένα από τα θέματα τα οποία ενδιαφέρουν ιδιαίτερα την Vivian Redding. Μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι μαζί οι δυο μας θα δώσουμε τη δυνατότητα αυτή να αντιμετωπίσουμε αυτό το ζήτημα. Δεν μπορούμε να αποδεχτούμε σαν δεδομένη αυτή την κατάσταση. Μια συμπληρωματική ερώτηση. Πιστεύετε ότι θα ήταν πρόσφορο να προχωρήσουμε σε μια ενδελεχή έρευνα για να εξασφαλίσουμε ότι η τωρινή νομοθεσία πράγματι μπορεί να διατηρήσει τα δικαιώματα των πολιτών. Ας παρακολουθήσουμε αυτή την κατάσταση. Προτού πάρουμε την οποιαδήποτε απόφαση, ας δούμε αν υπάρχει ακόμα πρόβλημα και εάν μπορεί να επιληθεί με άλλο τρόπο εκτός από νομοθετικές ρυθμίσεις. Αλλά προφανώς αυτό ενδιαφέρει ιδιαίτερα και την Βιβιάν Ρενδίνγκ. Σας ευχαριστώ, ο συνάδελφος Γκρίτσπ. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμη Επίτροπε, υποψήφια Επίτροπε, Νομίζω ότι αυτό το χαρτοφυλάκιο, όπως όλα τα άλλα, θα πρέπει να συνάδει με δύο βασικές αρχές, με την επικουρικότητα και την βιώσιμη ανάπτυξη. Λόγω του πεδίου εφαρμογής του χαρτοφυλακίου της ε, ψηφιακής ατζέντα. Να σας ρωτήσω λοιπόν, πώς οραματίζεστε την βιώσιμη ανάπτυξη σε ό,τι αφορά την πρόσβαση στο εμπριζωνικό διαδίκτυο, ιδιαίτερα σε απομακρυσμένες περιοχές, στην Ήπεθρο. Επίσης υπάρχει, υπάρχουν μεγάλες διαφορές μεταξύ των κρατών μελών, γιατί η πρόσβαση στο διαδίκτυο είναι πραγματικά πολύ διαφορετική και συχνά γίνεται και με παραδοσιακά δίκτυα. Τι θα αποδεχτείτε λοιπόν και πώς σκοπεύετε να προωθήσετε την εξέλιξη αυτή η απάντηση με τις τελευταίες κατευθυντήριες γραμμές για την ευρυζωνικότητα. Νομίζω ότι έχουμε δώσει μια σαφή απάντηση. Θα πρέπει να έχουμε ίσως πιο τακτικές επαφές και ενημέρωση των κρατών μελών. Αλλά αν θέλουμε πραγματικά να ακολουθήσουμε τη γραμμή αυτή της Επιτροπής, προκειμένου μέχρι το 2013 να υπάρχει 100% κάλυψη ευρυζωνική. Έχουμε ακόμα πάρα πολλά να κάνουμε. Και οι οικονομικές πτυχές του θέματος θα μπορούσαν να επιληθούν μέσα από τα κονδύλια τα οποία είναι διαθέσιμα, τα οποία θεωρώ ότι είναι ευρέως γνωστά, αλλά φυσικά θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν και ως τώρα το Κοινοβούλιο έχει μετανιώσει το ότι δεν έχει χρησιμοποιήσει αυτό το υψηλότερο επίπεδο που είχε προταθεί από τα κράτη-μέλη, αλλά σε κάθε περίπτωση βρισκόμαστε σε μια φάση επιτάχυνσης για να καλύψουμε τα κενά. Φυσικά, μέσω της ανακοίνωσης ο κόσμος θα πρέπει να ενημερώνεται και αυτό θα μπορούσε να γίνει μέσω της βιωσιμότητας, αλλά και μέσω άλλων ζητημάτων, όχι μόνο μέσω του ηλεκτρονικού εμπορίου, αλλά μέσω της ηλεκτρονικής υγείας, της ηλεκτρονικής εκπαίδευσης και ούτω καθεξής. Πολλά τέτοια θέματα. Και αυτό που μου είπαν πολλά κράτη-μέλη είναι ότι ενδιαφέρονται για μια συνεργασία και σε αυτόν τον τομέα. Να σας ρωτήσω Επίσης, κάτι αναφορικά με, τα, με τις γραπτές σας απαντήσεις. Το πρόγραμμα το οποίο αναφέρεται για την ηλεκτρονική υγεία, θεωρείτε ότι το πρόγραμμα αυτό θα μειώσει και τις πολιτισμικές διαφορές, τις διαφορές ως προς την εξέλιξη, την ανάπτυξη. Απάντηση. Ειλικρινά ελπίζω ότι με το πρόγραμμα που καλύπτει την ηλεκτρονική υγεία, που δεν γνωρίζει σύνορα, όντως θα χρησιμοποιηθούν και θα αξιοποιηθούν οι ευκαιρίες διασυνοριακής ε, παροχής τέτοιων υπηρεσιών. Και ίσως το αναφέρομαι υπερβολικά συχνά στην Δανία, αλλά αν καταφέρουμε να σημειώσουμε επιτυχία σε τέτοιου είδους προγράμματα, θα πετύχουμε με ένα σπάρο δύο τριγώνια. Θα λύσουμε δύο προβλήματα με μιας. Για παράλληλα, σε ό,τι αφορά τους ηλικιωμένους, θα λάβουν την υγειονομική περίθαλψη που χρειάζονται, θα τους δοθεί η ευκαιρία να ζουν αυτόνομα, αλλά παράλληλα θα έχουν και την ευκαιρία να λαμβάνουν τις υπηρεσίες αυτές σε χαμηλότερο κόστος. Και αυτό αποδείχτηκε μέσα από το παράδειγμα της Δανία. και ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά και την Ήπεθρο για παράδειγμα. Άρα τα παραδείγματα αυτά μας εμπνέουν. Θα πρέπει να μάθουμε ένα από τον άλλον. Και χάρηκα και ήμουν ιδιαίτερα περήφανη που είδα ότι η Δανία πλέον αποτελεί χώρο υπόδειγμα. Και είπα πλέον εξετάζει με βάση την δανεία πώς μπορεί να μιμηθεί το σύστημά της. Ας προσπαθήσουμε λοιπόν να υπάρξει αυτός ο σύνδεσμος με την ενιαία αγορά στην Ευρώπη. Από την Ο κύριος Σουάμπ. Ευχαριστώ κυρία Επίτροπε. Έχω μεγάλο σεβασμό για το έργο σας στην προηγούμενη θητεία. Είχατε σταθεί πραγματικά πολύ σκληροί πολλές φορές όπως πρέπει. Θα ήθελα όμως να σταθώ σε ένα σημείο το οποίο πρέπει να το αντιμετωπίσουμε λιγάκι πιο συγκεκριμένα. Ο κύριος Ρούμπικ αναγκάστηκε να φύγει. Ήθελα όμως να επανέλθω και να σας ρωτήσω τι θα κάνετε με, για την ε, οδηγία Roaming 2. <clears throat> τι ακριβώς θα κάνετε αν ο κανονισμός αυτός ο οποίος έχει εγκριθεί δεν φέρει τα αποτελέσματα τα οποία περιμένουμε προς όφελος του καταναλωτή. Θα προτείνετε ένα νέο νομοθέτημα ή όχι. Ένα νέο κανονισμό ή όχι. Αυτό το οποίο πρέπει να γνωρίζετε είναι ότι εγώ ενδιαφέρομαι πάρα πολύ για τα αποτελέσματα των συμφωνιών που έχουμε συνάψει. Οι συμφωνίες ήταν μεταξύ ημών με Y, της Κομισιόν και του καταναλωτή και των εταιριών φυσικά. Και αυτό φυσικά υποστηρίχθηκε από όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές και συγκεκριμένα τους παρόχους υπηρεσιών. Αυτό το οποίο πρέπει να είναι σαφέ είναι ότι δεν πρέπει να χωρεί καμία παρεξήγηση. Εάν δεν λειτουργήσει αυτή η συμφωνία, πάβει να υφίσταται. Και ξαναγυρίζουμε, τότε δεν θα ξαναγυρίσουμε βέβαια στο μηδέν. Εάν έχει νόημα λοιπόν αυτή η ρύθμιση, θα την υποστηρίξουμε. Δεν πρέπει να παραμείνει για πάντα αυτή η συμφωνία της περιαγωγής. Θα πρέπει να καταλάβουν όλες οι πλευρές ότι σε μια ανταγωνιστική αγορά μπορεί κανείς να έχει κερδοφορία, αλλά με τον τρόπο αυτό μπορούν να καρποφορούν και οι επενδύσεις. Αυτό ακριβώς ήθελα να τονίσω. Θα πρέπει να υπάρχει μια δυνατότητα <clears throat> να καταβάλει ο καταναλωτής ένα τίμημα το οποίο περιλαμβάνει και ένα πρόσθετο τίμημα που καλύπτει τον κίνδυνο. Αυτό είναι φυσιολογικό σε μια αγορά ζήτησης και προσφοράς. Αν το κατανοήσουν αυτό λοιπόν όλοι, εγώ νομίζω ότι θα γίνει κατανοητό ότι δεν σημαίνει ότι επειδή άλλαξε ο Επίτροπος για τα θέματα αυτά μπορούμε να επανέλθουμε στο παρελθόν. Ερμηνεύω αυτά που είπατε ότι είναι περισσότερο ναι από όχι. Αλλά τότε το δεύτερο ερώτημα μου είναι πιστεύετε τι θέλετε εσείς να ζητήσετε από τους ε, ε, ρυθμιστές, τους εθνικούς, με ποιο τρόπο θα μπορέσουν να, τι οδηγίες θα τους δώσετε για να μπορέσουν να φέρουν <clears throat> αυτή την αγορά στην κατάσταση που επιθυμείτε. Ποιε θα είναι, ποια θα είναι τα εγχειρήματα στα οποία θα πρέπει να προχωρήσουν. Μονάχα θέλω να τονίσω ότι είναι απαραίτητη η εμπιστοσύνη. Μόνο όταν κάποιος λέει ότι δεν δείχνει σημάδια ότι δεν μπορεί να τύχει εμπιστοσύνη, τότε μπορούμε να έχουμε μια διαφορετική αντιμετώπιση. Αν υπάρχει χάρη επίπεδο τιμών το οποίο δεν είναι αποδεκτό σε διάφορες κατηγορίες υπηρεσιών, μόνο τότε θα πρέπει να δράσει κανείς. Και νομίζω ότι τελικά οι εμπλεκόμενες πλευρές δεν κατανόησαν ή κατανόησαν και δεν ήταν έτοιμες να δράσουν. Αυτό έχει αντιμετωπιστεί ήδη δύο φορές. Νομίζω ότι όλες οι εμπλεκόμενες πλευρές θα πρέπει να την χάνουν καταρχήν της εμπιστοσύνης της Κομισιόν, να θεωρούμε ότι έχουν λάβει το σωστό μήνυμα και ότι εμείς είμαστε και εμείς σταθεροί στην δική μας στάση ως Κομισιόν. Αλλά καταρχήν θα πρέπει να δοκιμάσουμε την προσέγγιση η οποία έχει συμφωνηθεί και μόνο εάν δεν επιτύχει θα πρέπει να την αναθεωρήσουμε και έχουμε να περιμένουμε την ενδιάμεση αξιολόγηση και την τελική αξιολόγηση που θα δείξει ποιο ήταν το αποτέλεσμα αυτού του εγχείρηματο λήψη απόφαση. Θα έχουμε καιρό λοιπόν για να έρθουμε και πάλι σε επικοινωνία με τι εμπλεκόμενε πλευρέ. Ευχαριστώ για την Νομική Επιτροπή, η κυρία Γκάλο. Σας Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. κυρίε Υποψήφια Επίτροπε, θέλω να θέσω ένα ερώτημα εν ονόματι της Επιτροπής Νομικών Υποθέσεων που εκπροσωπώ εδώ και με την οποία σίγουρα θα πρέπει να συνεργαστείτε σε κάποια βασικά θέματα. Την εποχή της ψηφιοποίησης, ποια θα είναι τα βασικά σημεία της στρατηγικής σας που θέλει να δημιουργήσει ενιαία αγορά ψηφιακή για το δημιουργικό περιεχόμενο διατίθεται απευθείας online και τι πρόταση νομοθετική ε, έχετε υπόψη σας σε αυτό το πλαίσιο. Βλέπετε να υπάρχει κάποια ανάγκη να εφαρμοστεί η ευθύνη του τομέα, όπως στις τηλεπικοινωνίες, η ε, πάροχοι υπηρεσιών στο διαδίκτυο, πρόσβαση στο διαδίκτυο, εκείνων που χρησιμοποιούν παράνομα δημιουργικά ε, προϊόντα στο διαδίκτυο που προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα. Anyhow, um, Το παράνομο, η παρανομία δεν είναι αποδεκτή. Εν γέννη. Η παρανομία δεν είναι δεκτή. Αν υπάρχει η παραβίαση, αν δεν υπάρχει μόρφωση με τους κανόνες. Μιλώντας για τη δημιουργικότητα, εκεί πρέπει να ίσως να τα πάρουμε τα πράγματα πιο σοβαρά. Σε μια δημιουργική αγορά αγορά δημιουργίας, πρέπει να υπάρχει ισορροπία μεταξύ προσφοράς και τιμήματος που καταβάλλεται. Στις περισσότερες περιπτώσεις θα πρέπει να ακολουθείτε νομική, νόμιμη προσέγγιση μάλλον και νομική παρέμβαση αν υπάρχει παρανομία. Σε στενή συνεργασία πρέπει να κινηθούμε. και να λάβουμε ότι τα περισσότερα μέρη τα εμπλεκόμενα είναι κατά της υπερβολικής ρυθμίσεως. Αν όμως χρειάζεται και βελτιώνει τη διαφάνεια και τη σαφήνεια, τότε θα πρέπει να κάνουμε κάτι. Συμπληρωματική ερώτηση, κυρία συνάδελφε. Ευχαριστώ. Άλλο ερώτημα, πολύ συγκεκριμένο. Ποια είναι τα μέσα χρηματοδοτήσεως που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για να αναπτύξετε την Ευρωπαϊκή και σε αυτά τα πλαίσια. Σε συμφωνία υπάρχει δυνατότητα, πιθανότητα συμφωνίας με το Google. Απάντηση. Θα ήμουν κατά. Θα ήταν κατά των κανόνων πριν διότι και το Google δραστηριοποιείται σε αυτή την αγορά. Και πιστεύω στον ανταγωνισμό. Αυτό είναι κάτι που συντηρεί όλα τα εμπλεκόμενα μέρη, τα κρατάει ξύπνια. Ανθρώπους, εταιρείε, όλους. Είναι μια μεγάλη πρωτοβουλία η Ευρωπαϊκή. Είναι στην απαρχή της ασχολείται με το παρελθόν μας, με την ιστορία μας και έγκαιρα θα έλεγα και πρέπει να συνεχίσουμε. Να ασχοληθούμε με τις άλλες πτυχές. Δεν είναι μόνο τα ορφανά έργα και είναι και το θέμα ξανά της πνευματικής ιδιοκτησίας. Ας το πω θετικά. Βλέπω σαν πρόκληση το ότι το Google δραστηριοποιείται σε αυτόν τον τομέα και θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι αυτό σημαίνει αγγλική γλώσσα. Και αν θέλουμε να τηρήσουμε την κουλτούρα όλων των διαφορετικών γλωσσών μας σε αυτούς τους τομείς πολιτισμού και ιστορίας, θα πρέπει να σπάσουμε τον κύκλο. Διαφορετικά θα μας ξεπεράσουν σε κάποιε δραστηριότητε και πρωτοβουλίε και δεν μπορούμε να του κατηγορήσουμε διότι είναι ένα μέρο, συμμετέχουν στην αγορά. Θα πρέπει η Ευρωπαϊκή να μείνει στην προσοχή μα. Και θα πρέπει να συζητήσουμε με άλλα μέρη και να δείξουμε ότι δεν δεχόμαστε ότι η Ευρωπαϊκή θα μείνει ω έχει τώρα. Είναι καλή τώρα, αλλά θα πρέπει να ανοίξει τα φτερά τη. Κολέγιο Ο Κυρία Επίτροπε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πολύ καλές απαντήσεις που μας έχετε δώσει ως τώρα. Τα ψηφιακά μέσα επηρεάζουν με τεράστιο τρόπο το συνολικό τοπίο των μέσων, γιατί ο κόσμος θέλει όλο και πιο πολύ να διαβάζει online και δεν θέλει να πληρώνει συνδρομές. Το θέμα είναι τα έσοδα τα διαφημιστικά, τα οποία τα ρυθμίζουμε όλο και πιο πολύ στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Παρά το γεγονός ότι πρόκειται για μία ένδειξη της ελευθερίας έκφρασης. Και άλλο ένα πρόβλημα είναι ότι ένα μεγάλο μέρος των διαφημίσεων ε, online είναι στα χέρια της Google, πάνω από 50%. Άρα σας ρωτώ, θεωρείτε ότι αυτό διακυβεύει τον πληραλισμό των μέσων, γιατί αν δεν υπάρχουν έσοδα, δεν θα μπορέσουν να παράγουν τα σχετικά περιεχόμενα. Και αν υπάρχει τους κίνδυνους, τι σκοπεύετε να κάνετε. Απάντηση. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να συνειδητοποιούμε ότι δεν τίθεται θέμα. του κατά πόσο είμαστε υπέρ ή όχι. Ο πλουραλισμός των μέσων είναι κάτι το ευάλωτο στο οποίο μπορούν να επιτεθούν πολύ διαφορετικοί παράγοντες. Αυτό να το έχουμε υπόψη μας. Γι' αυτό λοιπόν συνδέεται και τόσο πολύ με την ελευθερία της έκφρασης και με τον πολιτισμό μας, τη δημοκρατία μας. Μπορώ να σας επαναλάβω την διακήρυξη, τη δήλωση που εγκρίθηκε τον περασμένο Οκτώβριο για την ελευθερία έκφρασης και ενημέρωσης πληροφόρησης στο Κοινοβούλιο αυτό. Αυτό που με εμπνέει είναι ότι φυσικά μετά από τις εμπειρίες μας με την Κίνα, τουλάχιστον αυτά που διαβάζουμε, όντως πρέπει να υπάρχει ισορροπία μεταξύ ελευθερίας έκφρασης και άλλων τέτοιων θεμελιωδών αξιών, όπως η προστασία για παράδειγμα των ανηλίκων και η ανθρώπινη αξιοπρέπεια, γιατί και αυτό φυσικά αποτελεί μια συνιστόσα στην όλη συζήτηση. Και αυτό θεωρώ ότι σημαίνει ότι πρέπει να υπάρχει νομοθεσία για την προστασία των ενηλίκων, της ιδιωτικής σφαίρας. Η καταπολέμηση των παράνομων περιεχομένων θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται στις προτεραιότητές μας και θα πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι σαφώς θα πρέπει να τεθούν τα θέματα αυτά, αλλά θεωρώ ότι ο πλουραλισμός των μέσων αποτελεί κάτι το απόλυτα θετικό, το οποίο θα πρέπει να προστατεύουμε. Δεύτερη ερώτηση. Χαίρομαι που στη συζήτηση για την απαγόρευση, που θα γίνει συζήτηση για την απαγόρευση των διαφημίσεων, είπατε ότι τα online περιεχόμενα και οι πληροφορίε online χρησιμοποιούνται όλο και πιο πολύ, αλλά και σε ευαίσθητου τομεί τη ζωή, όπω για παράδειγμα στην υγεία. Και βλέπουμε λοιπόν το εξή φαινόμενο, ότι ο κόσμος προσπαθεί να μάθει όλο και πιο πολλά πράγματα μέσα του διαδικτύου για την υγεία του και για φάρμακα και καταλήγει σε λάθος ε, πληροφορίες. Η κυρία Ρέντινγκ μιλούσε, είχε ξεκινήσει μια πρωτοβουλία για τις ε, πηγές που μπορεί κανείς να εμπιστευτεί κανείς. Ε, σκοπεύετε να συνεχίσετε αυτή την πρωτοβουλία. Απάντηση. Είναι σημαντικό. Είναι σημαντικό το γεγονός ότι δεν δεχόμαστε τα παραποιημένα προϊόντα. Όταν όμως μιλάμε για την υγεία, αυτά τα προϊόντα μπορεί να καταστούν άκρος επικίνδυνα και θα πρέπει λοιπόν να αναλάβουμε δράση. Ευχαριστώ ο συνάδελφος Ιβο Μπελέτ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κυρία Κρούς. Μετά από μία ώρα να σας κάνω και πάλι μία ερώτηση στα Ολλανδικά για να απαντήσετε στη μητρική σας γλώσσα. Ο συνάδελφος Χατζημαρκάκης μίλησε για τα περιεχόμενα online. Θα ήθελα να προχωρήσω λίγο παραπέρα. Όποιος θέλει αποτελεσματική προστασία των ε, ε, πνευματικών δικαιωμάτων και μία από τις δυνατότητες που έχουμε για την κατεύθυνση αυτή είναι ένα τέλος στους ψηφιακούς φορείς και στα διαδικτυακά, στις διαδικτυακές συνδρομές. Ξέρω ότι δεν είσαστε υπέρ των τελών αυτών, αλλά ίσως το μη χείρον βέλτιστο. Σας ε, ρωτώ λοιπόν ποια είναι η στάση σας απέναντι σε μια τέτοια προοπτική. Απάντηση. Είμαι διστακτική. Συμφωνώ μαζί σας μεν ότι θα μπορούσε να αποτελέσει ένα τμήμα της λύσης και αυτό σημαίνει ότι για μένα υπάρχει αυτή η τάση. Θα μπορούσε να σκεφτεί κανείς γιατί να μην ακολουθήσουμε αυτή την κατεύθυνση. Αλλά αφετέρου θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι τέτοιες, ε, τέτοια τέλη θα πρέπει να ρυθμιστούν. Σε κάθε περίπτωση μπορούμε να αναλογιστούμε αυτή τη δυνατότητα, γιατί σίγουρα αποτελεί μια σοβαρή λύση. Συμπληρωματική ερώτηση. Πολύ ενδιαφέρον αυτό που μόλις είπατε και σίγουρα θα το συζητήσουμε και περαιτέρω τους επόμενους μήνες. Άλλη μια ερώτηση. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει καταστήσει σαφές ότι δεν θέλει να εξαιρεθούν οι χρήστες του διαδικτύου, να τους κλειστεί η πρόσβαση στο διαδικτύο λόγω παράνομου κατεβάσματος. Και μιλήσαμε για μία για μια προσέγγιση ε, σε επίπεδα, για τη δηλαδή ενδεχομένως το να περιοριστεί η πρόσβαση στο ίντερνετ ανάλογα με τον όγκο που κατεβάζει ο καταναλωτής. Ποια είναι η στάση σας απέναντι σε αυτή τη λύση. Είστε πολύ δημιουργικός, αλλά αυτό το γνώριζα ήδη. Και εγώ και πολλοί άλλοι. Το πρώτο θέμα είναι το εξή. Τη συζήτησή σας για το πλαίσιο αυτό την παρακολούθησα και διαπίστωσα ότι βρέθηκε μια λύση με την ε, τροπολογία 183. Αυτή η τροπολογία θεωρώ ότι περιλαμβάνει βασικά, θεμελιώδη στοιχεία, τα οποία είναι πάρα πολύ σημαντικά και τα οποία σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να διασφαλίσουν την τήρηση της νομοθεσίας. Τώρα, το πώς θα μπορούσαμε να, διαμορφώσουμε τη δική σας πρόταση. Υπάρχει ο κανονικός, αν θέλετε, τρόπος και να λέμε ότι δεν θα πρέπει να γίνουν σφάλματα, αλλά υπάρχει ένας καλός τρόπος συνδυασμού με την τροπολογία 183 και αυτό θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Εκτός μικροφώνου η υπόλοιπη απάντηση. Σε πρώτη φάση, εκ πρώτη όψεως θα έλεγα ότι θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Προτού εισάγουμε μια τέτοια ρύθμιση, θεώρησα ότι η έκκληση που απευθύνατε με την τροπολογία και τον 83 ήταν πάρα πολύ σαφής. Ξέρω πόσο αίμα, δάκρυα και τρώτα κόστισε και σε ό,τι αφορά τη συζήτηση με το Συμβούλιο. Θεωρώ ότι βρισκόμαστε σε πολύ ευαίσθητο έδαφος. Ευχαριστώ κύριος Ματίας Γκρότ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κυρία Κρούς, έχετε μιλήσει για τον ανταγωνισμό μεταξύ των επιχειρήσεων προς το καλό των καταναλωτών. Από την 1η Δεκεμβρίου έχει τεθεί σε εφαρμογή η συνθήκη τη Λισαβόνα και εμεί έχουμε τονίσει αυτή τη συνθήκη εχετε θεσει ό,τι αφορά την ηλεκτρονική συμμετοχή των πολιτών. Γι' αυτό θα ήθελα να εχει μεγαλυτερη συμμετοχη ο πολιτη στι διαδικασιε ληψης αποφαση στην ευρωπαικη ενωση η ευρωπαικη επιτροπη εχει κανει πολλα περσι σε οτι αφορα την ηλεκτρονικη συμμετοχη των πολιτων γι αυτο θα ηθελα να ενδιαφερθω για το γεγονός για τις δραστηριότητε μάλλον που εσείς θα αναπτύξετε για να συνεχιστεί αυτή η στρατηγική της ηλεκτρονικής συμμετοχής για να γίνει πιο ανοιχτή η Ευρώπη και να μην μείνουν τόσα πολλά ερωτηματικά όσο αυτό που φοράτε σε σχέση με την ευρωπαϊκή πολιτική και να υπάρξει μεγαλύτερο ανοιχτό πνεύμα, περισσότερο ανοιχτό πνεύμα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Συμφωνώ απόλυτα θα πρέπει να συνεχίσουμε με την ίδια πορεία που είχαμε στο παρελθόν. Προσπαθώ να βρω την ε, μετάφραση του. Ε, του θαυμαστικού. Του... Θα μπορούσε αυτό ίσως να απαντήσει στο ερώτημά σας. Το ένα θαυμαστικό. Σαν σήμα. Συγκεκριμένα, στον τομέα αυτό τι θα αναλάβετε να πράξετε για την καλύτερη ε, συμμετοχή των πολιτών και επίσης στην αναγνωσιμότητα των στοιχείων που δίδονται μέσα από αυτήν την ε, συμμετοχή στα θεσμικά όργανα. Τι θα κάνετε λοιπόν συγκεκριμένα για να πείσετε τους πολίτες να συμμετέχουν περισσότερο και να ε, έχουν μια παρουσία. Όταν εμείς ε, ανακοινώσαμε ότι θέλουμε 100% ευζωνική κάλυψη, ότι θα εφαρμοστεί αυτό το μέτρο και θέσαμε το 2013 σαν καταληκτική ημερομηνία, θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ σαφείς έναντι των δυνητικών καταναλωτών, των ε, ενδιαφερομένων καταναλωτών σε σχέση με το τι θα γίνει. Αλλιώς είναι μια μονάχα μονόδρομη πληροφόρηση. Πρέπει να ξέρουν όλοι οι πολίτες ότι υπάρχει αυτή η απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να ξέρουν τι συνέπειες μπορούν να προέλθουν για τη ζωή τους, ότι αυτό μπορεί να είναι και ένα πολύ σημαντικό στοιχείο της σύνδεσής τους με το διαδίκτυο στον επαγγελματικό και ιδιωτικό χώρο, ότι θα αλλάξει τη ζωή τους. Για αυτούς οι οποίοι δεν το ξέρουν θα αλλάξει η ζωή τους. Η κυρία Νίμπλερ έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κυρία Υποψήφια Επίτροπε, Έχω παρακολουθήσει με μεγάλο ενδιαφέρον αυτή τη συζήτηση και σίγουρα υπάρχουν πολλά ερωτήματα τα οποία δεν έχουν τύχει απαντήσεως για το αν θα υπάρξει ρύθμιση νομοθετική για, το, για την περιαγωγή, αν δεν λειτουργήσει η αγορά. Αυτό έμεινε αναπάντητο αυτό το θέμα. Τι ακριβώς θα κάνετε για να εξασφαλίσετε την ουδετερότητα του διαδικτύου. Τι θα γίνει και σε διεθνές επίπεδο για το πακέτο τηλεπικοινωνιών το οποίο εμείς έχουμε ε, με μεγάλη δυσκολία εγκρίνει πώς θα προστατεύσετε την ελευθερία έκφραση στο διαδίκτυο, τι θα γίνει με την πολιτική ραδιοσυχνοτήτων. Για όλα αυτά τα θέματα δεν έχουμε ακούσει κάποια <clears throat> απάντηση. Δεν έχω την εντύπωση λοιπόν ότι σταθήκατε σαφείς για τα θέματα αυτά. Και θέλω να θέσω ένα ερώτημα. ποια θα είναι τα συγκεκριμένα μέτρα και τα κίνητρα τα οποία θα δώσετε για να υπάρξει αυτό το σημαντικό βήμα για την ευρωζωνική κάλυψη στην Ευρώπη, για να υπάρξει συνολική ευρωζωνική κάλυψη. Φαίνεται ότι υπάρχει μεγάλη παρεξήγηση όταν μιλάμε για την περιαγωγή το roaming. Ε, είχαμε επικοινωνήσει πάνω σε αυτό. Με τη Vivian Redding είχατε επικοινωνήσει. Πρέπει να γίνει διάμεση αναθεώρηση το καλοκαίρι φέτος και ένα χρόνο αργότερα θα γίνει η τελική έκθεση και αυτό που έμαθα ήταν ότι όταν ζητάς για μία έκθεση τα πορίσματά της αφορούν, κατα... αν είναι αρνητικά, βλέπεις αν η πολιτική σου πρέπει να αλλάξει, τι πρέπει να αλλάξει κλπ. Αυτό θέλω να πω. Αν λέω ότι το roaming 3 θα υπάρξει. Δεν περιμένω ότι θα λάβουν τα διάφορα εμπλεκόμενα μέρη, τα διάφορα μηνύματά μας. Έχουμε να κάνουμε με στοιχεία, δεδομένα, με μηνύματα, με SMS. Δεν είναι ξεκάθαρο το καλοκαίρι του 2011 ποιο θα είναι το τελικό αποτέλεσμα των αποφάσεων που λάβατε εσείς και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τούτου λεχθέντος. Δεν μπορείτε να μου ζητάτε να ανακοινώσω το roaming 3 για την περιαγωγή. Ε, που δεν είναι, δεν μπορεί να γίνει αυτό. Είμαι θετική από τη στιγμή που το πόρισμα θα με κάνει να αλλάξω γνώμη. Είναι ξεκάθαρα. Εάν δεν πρέπει να γίνει κάτι, εάν έχει γίνει κάποια παράβαση θα κάνω ό,τι πρέπει. Ουδετερότητα του δικτύου. Υπάρχει μόνο μία απάντηση. Ναι, είμαι ένθερμα υπέρ. Και ανέφερα το μικρό μηναματάκι. Έβαλα μία καρδούλα στην ουδετερότητα του δικτύου. Είναι αγαπημένο μου θέμα. Λοιπόν, τι διακυβεύεται εδώ για το περιεχόμενο στο διαδίκτυο online. Ελευθερία της έκφρασης. Εγώ είμαι υπέρ, κάθετα υπέρ. Θα σας εξέπλητα αν έλεγα το αντίθετο. Αλλά αυτό δεν μπορεί να γίνει χωρίς κάποια αντίδραση, αν το περιεχόμενο που διατίθεται δεν ταιριάζει με αυτά που θεωρούμε σωστά όσον αφορά την προστασία των ανηλίκων, και τι βλέπουν τα παιδιά στο διαδίκτυο ανήλικοι και αν είναι κατά τη αξιοπρέπεια το περιεχόμενο, τότε αν ισχύουν αυτά θα πρέπει να αντιδράσουμε σε αυτό το περιεχόμενο που διατίθεται online. Ευρυζωνική ε, σύνδεση είμαι υπέρ 100% και ξέρω ότι αναλαμβάνω ένα κίνδυνο όταν το λέω αυτό και όταν αναφέρομαι στο χρονοδιάγραμμα. Μπορείτε να με κατηγορήσετε να αργήσω έξι μήνες. Και αν με υποστηρίξετε εγώ αυτή τη θέση, θα μου χτυπήσετε την πόρτα και θα μου πείτε, έλα, έλα, έχεις γραπτή δήλωση ότι θα είσαι έτοιμη και υπέρ. Όχι μόνο υπέρ, ότι θα παρουσιάσεις κάτι που μπορεί να υποστηρίξουν 100%. Τον αναλαμβάνω τον κίνδυνο. Έχοντας πλήρη επίγνωση ότι αυτό είναι που χρειάζεται η Ευρώπη. Μία συμπληρωματική ερώτηση για την Συμπληρωματικό ερώτημα. Είχα θέσει ένα συγκεκριμένο ερώτημα. Τι γίνει αν οι αναλύσει δείξουν ότι δεν λειτουργούν οι ρυθμίσει σα. Είπατε ότι θα δράσετε. Τι σημαίνει αυτό θα, ότι θα δράσετε. Τι σημαίνει αυτό σε συγκεκριμένο επίπεδο. Και επίση για την υποδομή τον, την ευρωζωνική. Στην προηγούμενη απάντησή σας είπατε ότι έχετε κάνει αλλαγές στην οικονομία, έχετε ε, διαλύσει μεγάλους ομίλους και τα λοιπά, ως επίτροπος ε, ε, ανταγωνισμού έχετε κάνει σημαντικά πράγματα. Αυτό πρέπει να το παραδεχτώ. Τώρα, στην περίπτωση που δεν έχετε αυτά τα μέσα στη διάθεσή σας, με ποιο τρόπο θα εξασφαλίσετε ότι θα υπάρξει προώθηση της υποδομής για, την, για, την, για τα βρυζονικά. Πώς θα πείσετε τους μεγάλους διεθνείς παίκτες να επενδύσουν προς την κατεύθυνση αυτή. Φανταστείτε τα συμπεράσματα της ελίκης εκθέσεως του 2011 και φανταστείτε ότι τα, πορίσματα είναι καταστροφικά όσον αφορά την περιαγωγή. Εντελώς αρνητικά. Τότε τα εμπλεκόμενα μέρη στην αγορά θα πρέπει να ξέρουν θα δράσουμε και ίσως εκεί να βγει το roaming 3. 3. Είμαι θετική όμως εγώ. Οι προσδοκίες μου είναι θετικές. Βεβαίως εξαρτάται από τα απορίσματα της τελικής εκθέσεως. Ας πούμε ότι δεν είναι θετικά τα αποτελέσματα ή για κάποια, κάποιες πτυχές είναι αρνητικά τα πορίσματα. Θέλω να ξέρω πού έγκυται το πρόβλημα, ποια είναι η για καποια καποιες πτυχες ειναι αρνητικα τα απορισματα θελω να λύση και τι είδους λύση χρειαζόμαστε έναν τυπίου ούτως ώστε στο τέλος να βρούμε μια λύση που υποστηρίζουμε όλοι και ο καταναλωτής να πληρώνει για μια υπηρεσία, αλλά να μην είναι το τίμημα υπερβολικό. Να είναι κανονικό το τίμημα που καταβάλει ο καταναλωτής για την παρεχόμενη υπηρεσία. Συναρτήσει των πορισμάτων της εκθέσεως θα κινηθούμε. Αναφέρατε ότι Επίτροπος Ανταγωνισμού και ταυτόχρονα όντα, ότι είναι διαφορετική θέση του Επιτρόπου περί ανταγωνισμού με τη θέση του Επιτρόπου για το συγκεκριμένο χαρτοφυλάκιο που μου προτείνεται τώρα. Ε, δεν ασχολιόμαστε μόνο με ε, κυρώσεις και με διορθώσεις όταν ήμουν Επίτροπος Ανταγωνισμού. Προσπαθούσαμε να, να δημιουργήσουμε μέσα λύσεις, ε, επικοινωνία, να χτίσουμε γέφυρες για να βρούμε μια λύση. Και για να το κάνεις αυτό έχεις επιχειρήματα. Αν έχεις καλά επιχειρήματα, προχωράς. Και αν καταλάβει το άλλο μέρος το περιεχόμενο του επιχειρήματός σου, τότε μπορεί να καταλήξει σε κάποια λύση που είναι παραγωγική. Η συνάδελφη Μαρκής, κυρία Κρούς, τελευταία ερώτηση. Η, το η ομάδα των δημοκρατών ανησυχεί για το εξή. Για την κοινωνική πτυχή, το κοινωνικό σα όραμα, άκουμε που μιλάτε για επιχειρήσει, για ίσου όρου, μιλάτε για τεχνολογία, για κανόνε, αλλά δεν ακούω να μιλάτε για τον άνθρωπο, δεν ακούω να μιλάτε για τι θέσει εργασία και δεν ακούω να μιλάτε για τις τεράστιες δυνατότητες που θα, προ... θα... θα σημαίνει το χαρτοφυλάκιό σας για να ε, ξεπεράσουμε την οικονομική κρίση και μια δεύτερη εύκολη ερώτηση. Πότε θα θέσετε ένα τέλος στην ηγεμονία της Microsoft όπως το κάνατε και στην προηγούμενη σας ιδιότητα. Απάντηση. Έχω ένα πρόβλημα, κύριε Πρόεδρε. Αντιλαμβάνομαι απόλυτα, αλλά δεν μπορώ να το περάσω αντιλαμβάνομαι απόλυτα ότι στις αρχικές μου παρατηρήσεις αναφέρθηκα στο ότι αυτή η ψηφιακή ατζέντα θα είναι για τον καταναλωτή, για τον πολίτη στην Ευρώπη. Και αυτό αποτελεί τη βασική θέση κίνηση. Το επόμενο βήμα που έκανα ήταν να επιδείξω τα διάφορα θέματα τα οποία θα πρέπει να λάβουμε υπόψη για να μεταφράσουμε αυτή την πολιτική σε πράξεις, σε δράσεις για τον, για τον καταναλωτή, μιλώντας για την ηλεκτρονική υγεία. Αναφέρθηκα ίσως υπερβολικά πολλές φορές στο παράδειγμα της Δανίας, αλλά όντως πρόκειται για ένα από τα θέματα τα οποία με απασχολούν. Μίλησα για τους ηλικιωμένου. είπα ότι θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι αυτό θα μπορούσε να σημαίνει πάρα πολλά για τα ηλικιωμένα άτομα, τα οποία προτιμούν στις πιο πολλές περιπτώσεις να ζουν αυτόνομα όχι να μπουν σε κάποιον οίκο ευγυρίας. Πρόκειται λοιπόν για ένα θέμα το οποίο θα πρέπει να προωθήσουμε. Και αν τίθεται θέμα υποδομής, θα πρέπει και αυτό να το αντιμετωπίσουμε. Μίλησα για την εκπαίδευση, μίλησα για, για τους ανηλίκους. Πρόεδρε. Πώς αλλιώς μπορώ να εξηγήσω αυτό που εννοώ. Για πολλά μπορείτε να με κατηγορήσετε, αλλά και στο χαρτοφυλάκι του ανταγωνισμού θεωρώ ότι σημείωσα επιτυχία γιατί κατάφερα να έρθω σε επαφή με τον κόσμο, στον δρόμο, στα μαγαζιά. Όταν ο κόσμος με ρωτούσε στην αρχή τι ακριβώς κάνω, τώρα πια ξέρουν ότι η πολιτική του ανταγωνισμού στην τελική ανάλυση ανάλυση τον καταναλωτή επηρεάζει. Για θέσει εργασία, ασφαλώ, για οικονομία μιλάμε, για θέσει εργασία μιλάμε. Τι άλλο. Αναφέρθηκα στι θέσει εργασία, αναφέρθηκα στις, στην οικονομία, στι μικρομεσαίε επιχειρήσει. Αισθάνομαι ελαφρώ ε, αδικημένη και λυπάμαι που δεν πέρασε αυτό το μήνυμα. Αλλά χαίρομαι για την παρέμβασή σας. Ελπίζω τώρα στην αρχή και στο τέλος της ακρόασης να κατάφερα να πω ότι η ψηφιακή ατζέντα στο σύνολό της αφορά τον κόσμο, αφορά τους όρους επί τους οποίους, από θα ήθελε να εκατομηθεί η Ευρώπη ο πολίτης. Άρα να θεωρήσω ότι θα εστιαστείτε στην πολιτική σας τον άνθρωπο και πρώτα απ' όλα στον άνθρωπο πριν και πάνω από όλες τις δυνατότητες για τις επιχειρήσεις. Φυσικά και όλα αυτά είναι πολύ σημαντικά, αλλά εμείς θέλουμε η προοπτική να είναι ο άνθρωπος και ο πολιτισμός. Και θα ήθελα να μου απαντήσετε και στη δεύτερη ερώτησή μου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Υπάρχει μία παρανόηση αν θεωρείτε ότι το να μιλάει και τις επιχειρήσεις δεν αφορά τον άνθρωπο. δεν είναι κάτι το αφηρημένο οι επιχειρήσει, δεν είναι κάτι που δεν αφορά θέσει εργασία, θέσει εργασίας αφορά, οικογένειε αφορά, που ζουν από τι επιχειρήσει από αυτές και εξαρτώνται από αυτές. Άρα, μπορείτε να θεωρήσετε ότι για μένα ο άνθρωπος είναι σε κεντρική θέση. Ιδάλλως δεν θα ήμουν στην πολιτική ζωή για την Microsoft. Μπορεί να, να είσαστε σίγουροι ότι και αυτό θα το αναλάβουμε εκ νέου, αλλά το κάναμε και την προηγούμενη περίοδο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν είναι δυνατόν να βγαίνουμε και να διακηρύττουμε πράγματα τα οποία τελικά δεν θα εφαρμόζουμε. Και στην περίπτωση της Microsoft μπορεί να είστε απόλυτα βέβαιοι ότι για τις ανοιχτές πηγές θα μείνουμε στο πλαίσιο των ε, θεσμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα καταβάλουμε κάθε προσπάθεια μάλιστα. Και έτσι λοιπόν ε, ακούσαμε όλες τις ερωτήσεις και όλες τις απαντήσεις λέει ο Πρόεδρος και όπως προβλέπετε και στη διαδικασία έχει καταλεκτικά πέντε λεπτά χρόνο η κυρία Κρούς για να κάνει τα σχόλιά της. Και στη συνέχεια θα ολοκληρώσουμε τη σημερινή ακρόαση. Έχετε το λόγο, κυρία Κρούς. Εκτιμώ ιδιαίτερα, κύριε Πρόεδρε, το γεγονός ότι μου δίνετε και πάλι το λόγο, γιατί θέλω να τονίσω ότι για να προωθήσουμε την ψηφιακή ατζέντα θα πρέπει να αναρωτηθούμε. Θέλω να ευχαριστώ λοιπόν τα, εσάς κύριε Πρόεδρε και την Επιτροπή Βιομηχανίας για τα ερωτήματά σας. Βρισκόμαστε σε ένα σταυροδρόμι χρειάζεται να βρούμε νέους τρόπους να εξασφαλίσουμε την οικονομική ανάπτυξη και αυτό για τους ανθρώπους μας. Οι επιχειρήσεις της Ευρώπης λοιπόν προσβλέπουν σε μας να κάνουμε τη ζωή τους λίγο καλύτερη και λίγο πιο εύκολη και ίσως και λίγο περισσότερο. Η ψηφιακή ατζέντα, γνωρίζετε, η ψηφιακή ατζέντα είναι το κλειδί σε αυτή την πρόοδο. Είναι τεράστια η πρόκληση, αλλά με την υποστήριξη και τη στενή συνεργασία με εσά, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και με την υποστήριξη του Προέδρου σας, μπορούμε να πετύχουμε σημαντικά πράγματα τα επόμενα πέντε χρόνια. Αν με επιβεβαιώσετε σαν Επίτροπο για την ψηφιακή ατζέντα, η αισιόδοξη Νέλη Κρούς θα εργαστεί για να βελτιώσει την κατάσταση επί τη βάση της ισχύως της Ευρώπης. Και η ρεαλιστική Νέλη Κρούς θα θυμάται ότι δεν μπορούμε να ξεκουραστούμε ούτε ένα λεπτό. Και αν με επιβεβαίωσετε, η πραγματιστική Νέλη Κρούς θα ακούσει τις απόψεις όλων αυτών που έχουν καλές ιδέες για να μπορέσουμε να προωθήσουμε την ατζέντα προς το εμπρός. Και θέλω να υπενθυμίσω τα έξι, τα έξι βασικά στοιχεία, δομικούς λήθους που ανέφερα έρευνα και καινοτομία, υποδομές, πρόσβαση και προσόντα, διαλειτουργικότητα και ανοιχτά στάνταρτ και η προγράσπιση της ενιαίας αγοράς. Αν δώσουμε έμφαση σε αυτά τα έξι θα μπορέσουμε να δώσουμε στην Ευρώπη την καλύτερη δυνατότητα να επιτύχει στις αγορές αυτές και αυτό θα βοηθήσει μια γενιά ε, να μεγαλώσει με οικονομική ανάπτυξη και θέσεις απασχόλησης. Πολλές φορές βλέπετε τα πράγματα όπως είναι και ρωτάτε γιατί είναι έτσι. Εγώ οραματίζομαι πράγματα που δεν υπήρξαν ποτέ και ρωτάω γιατί όχι κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, νομίζω ότι έχετε δίκιο όταν παραθέσατε αυτήν την ρίση. Αν με υποστηρίξετε μπορούμε να εξασφαλίσουμε την αλλαγή και ως πεπισμένη Ευρωπαία βασίζομαι στην υποστήριξή σας για να μπορέσουμε να προωθήσουμε τις ευκαιρίες και να φτάσουμε σε μια πραγματική ευρωπαϊκή ψυχιακή ατζέντα. Σας ευχαριστώ κυρία Κρούς για τις απαντήσεις σας, για τον χρόνο σας, για την παρουσία σας, για τη δέσμευσή σας. Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους που έθεσαν ερωτήματα. Έχουμε τελειώσει την ε, ακρόαση. Στις 8 θα συνεδριάσουν οι συντονιστές εκεί που έχουμε συμφωνήσει και για τους υπόλοιπους συναδέλφους τους εύχομαι καλό βράδυ.